Allora, riprendiamo la seduta. Intanto... Να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Dicevo, riprendiamo la seduta eh, pomeridiana. Mi scuso per il ritardo. Non... Να συνεχίσουμε λοιπόν με την απογευματινή συνεδρίαση. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Συνήθω δεν την καθυστερώ, αλλά μόλι τελείωσα μια συνάντηση με τον ε, Ιρλανδό Υπουργό Δικαιοσύνη για θέματα που αφορούν την Επιτροπή μα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με το απογευματινό τμήμα της συζήτησης. Εδώ έχουμε πληροφορίες, έρευνα και ε, προσαγωγή για απάτη ΦΠΑ. Έχουμε εδώ τον κύριο Φρανκ Φίλιψεν, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα θέματα καταπολέμησης για τα διασυνοριακά εγκλήματα και κατόπιν ο κύριος Ρέινο Νίλσεν, ο οποίος ε, είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος Καταπολέμησης της Απάτης και Πληροφοριών της Δανίας και θα μιλήσει για την καταπολέμηση του οργανωσμένου εγκλήματος για την απάτη ΦΠΑ και κατόπιν ο κύριος Τόμας Γκάιερ από τη Βόνη, από τη Γερμανία, που θα μας ε, μιλήσει για την έρευνα και τις, τη νομική δικαστική συνδρομή για την καταπολέμηση κατά της απάτης ΦΠΑ. Oh, Monsieur Philipsen, c'est le premier. nel dare la parola a Frank Phillips δίνω το λόγο στον Φρανκ Φίλιμσεν να σας πω όμως το εξή. Είχαμε ε, υπολογίσει αν ένα τέταρτο καθένας για να μιλήσετε. Λόγω όμως πίεσης χρόνου θα ήθελα να σας ζητήσω να περιοριστείτε στα 10 λεπτά. Πράγμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, προέρχομαι από την ειδική φορολογική επιθεώρηση εδώ πέρα στο Βέλγιο και η λέξη κλειδί όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, απάτης του ΦΠΑ, ειδικά στο διεθνή είναι συνεργασία, συνεργασία, συνεργασία. Είμαστε δύο που ασχολούμαστε με αυτόν τον ε, τομέα, εγώ και ο Γιάννικ Ιλό. Όσον αφορά λοιπόν την απάτη του ΦΠΑ, του λεγόμενο καρουσέλ, έχουμε μια παλιά ιστορία η οποία βεβαίως δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το οποίο είχαμε ε, και όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση ήταν όταν ξεκίνησε η Τελωνιακή Ένωση του Benelux και εκεί πέρα εμφανίστηκαν οι δυνατότητες της απάτης αυτή. Και βεβαίως το 1993 είχαμε την εισαγωγή του προσωρινού συστήματος όπου είχαμε μια εκρηκτική αύξηση ε, των κρουσμάτων αυτών και βλέπουμε πως ε, εμφανίστηκαν ε, ξανά από την δεκαετία του 70 κάποιες περιπτώσεις ξανά το 1998. Και συχνά βεβαίως ε, έχουμε περιπτώσεις ε, που βρίσκονται συνεχώς σε αντιπαράθεση με την αστυνομία, με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με ε, διάφορες αρχές. Οπότε έχουμε πάντα το ότι η απάτη καρουσέλ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για διάφορες ε, συμμορίες. Οπότε θα προσπαθήσω έτσι κάπως λογοτεχνικά να σας περιγράψω τι είναι αυτή η απάτη. Είναι ένα στρώμα, ένα... ένα ε, είναι ένας χήμαρος, με συγχωρείτε θα έλεγα, ε, τον οποίο εμείς προσπαθούμε να αδειάσουμε με κουβάδες και πρέπει συνεχώς αντί να αδειάζουμε κουβά-κουβά έναν χήμαρο, να φτιάξουμε κάποια φράγματα ή τις όχθες για να έχουμε δομές τέτοιες οι οποίες θα εμποδίσουν την ε, απάτη αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, για αυτό το οποίο ε, λέμε προληπτική διαχείριση του κινδύνου και προληπτική ανάλυση του κινδύνου. Και εμείς θεωρούμε πως είναι πολύ καλύτερο να αποφύγουμε εκ των προτέρων κάποια λάθη και ελλείψεις από το να προσπαθούμε εκ των υστέρων να τα διορθώνουμε. Και εδώ πέρα χρειάζεται η σωστή ε, προσέγγιση. Και εδώ πέρα ακριβώς χρειάζεται η στήριξη ε, της ευρωπαϊκής ε, ιδέας, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 904 του 2010. Βλέπετε, όπως είπα, πως ε, έχουμε αρκετές ε, εμπειρίες. Παλαιότερα προσπαθούσαμε να σχηματίσουμε και να διαγράψουμε πλήρως από το α έως το ω την πορεία της ε, απάτης. Τι γινόταν όμως, ενώ φτιάχναμε έναν υπέροχο φάκελο της όλης περίπτωσης, ήταν πάρα πολύ αργά όταν είχαμε ολοκληρώσει την υπόθεση. Οπότε έχουμε περάσει τώρα σε αυτό το οποίο βλέπετε στο δεξί μέρος του διαγράμματος. Δηλαδή κάνουμε μια γρήγορη ανείχνευση, μια έγκαιρη ανείχνευση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ε, απάτη ήδη πριν γίνει η πρώτη ε, αχρεώστητη πληρωμή να μπορέσουμε να τους ε, σταματήσουμε και αυτό. Βεβαίως σημαίνει πως δίνουμε μεγάλη σημασία σε όλα τα σημάδια που ε, καταδεικνύουν μια τέτοια απάτη γιατί βεβαίω αυτό συνδέεται με άλλες ε, απάτες στον τομέα της φορολογίας, των ειδικών φόρων, τελωνιακές απάτες κτλ. κτλ. Οπότε για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε αμέσως να σταματήσουμε αυτή την περίπτωση. Αν πάμε στο παρελθόν, βλέπετε εδώ πέρα τα επίσημα στοιχεία, παρατηρούν πως το 2001 είχαμε απώλειες στο Βέλγιο γύρω στο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω αυτής της απάτης. Κάτι το οποίο καταφέραμε να μειώσουμε. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2012 μιλούν για μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν να σκεφτούμε τις ε, διάφορες επιθεωρήσεις, τη συνεργασία με την εισαγγελία, με τα δικαστήρια, με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και βεβαίως την εκπαίδευση ε, εξειδικευμένων υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με τις διεθνείς δομές. Γιατί έχουμε την λεγόμενη ε, κλασική απάτη και το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα. Οπότε θα πρέπει να δούμε το εξής. Μαθαίνουν οι απατεώνες και διδάσκονται από κάθε αντιπαράθεση και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια σαφή ε, αντίληψη και όψη του φαινομένου. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έχουν μια άποψη, αλλά βεβαίως δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ορισμό για να μπορούν όλοι οι ελεγκτές, όλοι οι υπάλληλοι να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Οπότε βασική αρχή είναι να κάνουμε μια περιγραφή της τυπολογίας των διαφόρων μορφών με τις οποίες εμφανίζεται αυτή η απάτη. Κάποιες βεβαίω είναι πιο δημοφιλείς από άλλες, αλλά θα παρατηρήσετε εδώ πέρα στον χρωματιστό κύκλο από το 2000 μέχρι το 2003 έχουμε κατατάξει και τα ποσοστά των διαφόρων μορφών της απάτης. Έχουμε τα ψεύτικα τιμολόγια, τα κυκλικά τιμολόγια, τις ε, ψεύτικες ε, χρεώσεις και δαπάνες κτλ. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τον ίδιο ορισμό για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως είπα, να μιλούν την ίδια γλώσσα. Όσον αφορά την νομοθεσία, η νομοθεσία έχει εμπνευστεί από την ε, ευρωπαϊκή νομολογία Και βεβαίως μιλάμε και για καλύτερη διεθνή συνεργασία, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία εντός της ίδιας της χώρας, γιατί υπάρχει το πρόβλημα πως από χώρα σε χώρα διαφορετικές αρχές έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, άλλες έχουν δικαστικές και άλλες έχουν ε, αστυνομικές αρμοδιότητες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος της αντίδρασης. Επίσης, κάτι άλλο, θα πρέπει να είμαστε ε, πιο γρήγοροι και δραστήριοι από τους αντιπάλους μας που σε αυτή την περίπτωση είναι οι απατεώνες. Έχουμε λοιπόν την Eurofisk ε, η οποία συστάθηκε με τον γνωστό κανονισμό του 2010 και καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό καταπολέμησης απάτης, κατόπιν ορίσαμε την ομάδα εργασίας και ε, καταλήξαμε σε μία ομάδα πολυμερούς ανταλλαγής πληροφοριών και τέλος βεβαίως κάτι το οποίο είναι μια ελπίδα για εμάς, μια φιλοδοξία για εμάς να καταλήξουμε να κάνουμε μια κοινή ανάλυση κινδύνου μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Γιατί βεβαίως, όπως σας είπα, πρέπει να περάσουμε στην πρόληψη. Τέλος, θα κάνω μια σύνοψη και μετά τον λόγο θα πάρει ο συνάδελφος. Υπάρχουν τέσσερις α, ομάδες και τομείς εργασίας, το βλέπετε απάτη έμπτικ, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροπλάνα και τα λοιπά. Και το τρίτο τρίτος τομέας εργασίας είναι οι τελωνιακές ε, διαδικασίες και η απάτη ΦΠΑ. Και βεβαίως προσπαθούμε να παρατηρούμε σε πραγματικό χρόνο να ξέρουμε νέες ιδέες απάτης ε, για να τις προσθέσουμε στην λίστα του Καρισέλ. Η πρώτη, λοιπόν, ο πρώτος τομέας εργασίας γίνεται μέσω data mining και ε, διασταύρωσης ε, στοιχείων για να μπορέσουμε να δούμε διάφορες τάσεις οι οποίες εμφανίζονται. Οπότε τα πλεονεκτήματα του Eurofisk είναι πως έχουμε συνεργασία εξειδικευμένων ομάδων καταπολέμησης της απάτης, πως ε, ο κάθε ένας λοιπόν είναι εξειδικευμένος στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει η ταχύτητα υπάρχει ο αυθορμητισμός, είμαστε στοχευμένοι, είμαστε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού οράματος και επικρατεί και ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Και βεβαίως ε, αυτό είναι θετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρξε πρόοδος τα τελευταία χρόνια με το Ευρωφίσκ. Η αντίδραση των χωρών μελών οι αντιδράσεις ήταν διαφορετικές διστάζουν οι περισσότερες. Άλλες έχουν τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης του κινδύνου, άλλες θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στις αναλύσεις και το συνδυασμό των δεδομένων. Επίσης πρέπει να υπάρξει συνδυασμένη αντίδραση για τα, την ερμηνεία των στοιχείων για να μπορέσουμε να έχουμε μια σφαιρική άποψη. Εφόσον λοιπόν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών είναι και δικτών είναι ικανοποιητικό, υπάρχουν έγκαιροι δείκτες, το Eurofisk έχει το καλύτερο εργαλείο συλλογής και ανάλυσης τέτοιων στοιχείων και γι' αυτό πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνδυασμού, συντονισμού για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις αντιδράσεις μας, να βλέπουμε τις απάτες ε, συνολικά και να μπορούμε έτσι συνολικά να αντιδρούμε και από κοινού. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τη λεγόμενη Quick Analysis Team στο Eurofisk. Δηλαδή μια μονάδα για ακριβώς την ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων που να επιτρέπει αντίδραση η καταλληλότερη αντίδραση και ιδιαίτερα από κοινού. κοινού. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε κοινή αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις διότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στην καταπολέμηση των απατών. Όλα γίνονται μέσω του ίντερνετ, πολύ γρήγορα λοιπόν, άειλα και αυτό καμιά φορά ευνοεί τους απατεώνες. Όταν μιλάμε για διεθνοποίηση εννοούμε παγκοσμιοποίηση στην ουσία. Γιατί αυτό αφορά όλες τις χώρες του κόσμου με τη χρήση των πλασματικών τραπεζών που μπορούν να ιδρυθούν παντού. Επίσης πολύ επικίνδυνο φαινόμενο που μεγάλες εταιρείες καλής πίστεως όπως Καρουσέλ και εφαρμογή διαφόρων μονόπλευρων μονομερών ε, πρωτοβουλειών που τελικά δεν συμβάλλουν σε πολιτική εναρμόνιση. Γι' αυτό η πρόταση του Quick Reaction Mechanism θα μπορούσε να βλάψει τις δικές μας προσπάθειες. Προς στιγμή η Quick Reaction Mechanism καταλήγει σε μία αυτοκατάργηση, αυτο κατάσχεση δηλαδή εφόσον εφαρμοστούν πολλές εξαιρέσεις καταλήγουμε απλώς στη μετακίνηση της απάτης. Θέλουμε να δούμε όμως προς τα πού κινείται, προς ένα γενικευμένο σύστημα reverse charge. Αυτό κατ' εμένα θα αντιπροσώπευε ένα κόστος που ακόμη δεν το ξέρουμε και μεγάλη νομική ασάφεια και ο άχθος και για τις επιχειρήσεις. Και θα ήταν η παναχώρηση που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τα εθνικά ταμεία. Αυτά. Νομίζω λοιπόν τελικά ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Quick Analysis Team που σας έλεγα στα πλαίσια του Eurofisk. Η πρόταση αυτή θα γίνει τον Μάρτιο σε εσά. Ελπίζουμε να τη δεχτούν τα κράτη-μέλη τα περισσότερα και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα μέτρα της γενικευμένης αυτοκατάργησης για να μην μειωθούν έτσι τα έσοδα της Ένωσης με εθνικά μόνο κριτήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα για 10 λεπτά στον κύριο Ρέινο Νίλσεν. Ja, tak. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησαν οι συνάδελφοι. Όπως ε, ακούστηκε, και εμείς ασχολούμαστε με την απάτη καρουσέλ. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε επικεντρωθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Και σε κάποιο βαθμό έχουμε αφήσει στην άκρη το πιο παραδοσιακό μοντέλο απάτης η απάτη καρουσέλ εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε και τη σήμερα μέρα δεν είναι περιορισμένη απλώς και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει διευρυνθεί και αποτελεί πλέον ε, πρόβλημα διεθνούς απάτης. Υπήρχε και μία τάση βάσει της οποίας ε, παραδοσιακά προϊόντα, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, υπολογιστές, ε, ανταλλακτικά ε, κινητών τηλεφώνων και κινητών υπολογιστών, ενώ αυτά στην αρχή ήταν τα βασικά προϊόντα που ήταν αντικείμενο απάτης καρουζέλ, τώρα πλέον έχουμε επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα, ακόμα και σε παροχή υπηρεσιών και σε άειλα αγαθά. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε προσφάτως είναι ότι υπήρχε μαζική απάτη που σχετιζόταν με την εισαγωγή ενός συστήματος ε, ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών ε, στο εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και πρόκειται για ένα εικονικό σύστημα έπρεπε κάποιος να, κάνει, να είναι καταχωρημένο σε μια χώρα για να μπορεί λοιπόν να κάνει ανταλλαγή ε, εκπομπών και υπήρχε δυνατότητα να ε, γίνει σύνδεση με κάποιον ο οποίος προερχόταν από άλλη χώρα δεν υπήρχε ανάγκη για καταχώρηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούσε οποιοδήποτε να εγγραφεί στο Μητρό και από εκεί και πέρα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή εκπομπών και οι εκπομπές ε, ανταλλάσσονταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπήρξαν ε, σημαντικές απώλειες για τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω αυτής της μορφής απάτης. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς ακριβώς ε, σε ποιο βαθμό ε, έχει φτάσει αυτή η απάτη. Ε, οι έρευνες είναι εξελίξει, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Η Europol έκανε μια αξιολόγηση και εκτιμά ότι οι απώλειες είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, δεν ξέρω αν το σωστό ποσό είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι πρόκειται για πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία τέθησαν ήταν ότι δεν ήταν αρμόδιες οι φορολογικές αρχές, αλλά ε, τις πληροφορίες αυτές ε, τις έχουν άλλες αρχές και οι φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών δεν έχουν απαραίτητο πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ορισμένες φορές είναι οι αρχές ε, αρμόδιες για την ενέργεια που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον ενός συστήματος όπου οι ελεγκτικές αρχές, δηλαδή οι φορολογικές αρχές, δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, δεν υπάρχει διαφάνεια και επομένως δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την απάτη χωρίς να διαθέτουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Γεγονός το οποίο ε, επέτρεψε τελικώς αυτό το σύστημα να δημιουργηθεί αρχικώς και να εξελιχθεί στη συνέχεια. Ε, σήμερα πλέον οι κανόνες ανταλλαγής εκπομπών έχουν τροποποιηθεί, ευτυχώς, αλλά ε, χρειάστηκε αλλαγή της νομοθεσίας και τα κράτη-μέλη αντίδρασαν αρκετά γρήγορα, ιδίως μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι ε, τροποποιήθηκε η νομοθεσία και οι υποχρεώσεις ε, ε, των κρατών μελών και έτσι επιλύθηκε το πρόβλημα για τις χώρες οι οποίες είχαν εγκρίνει τους κανόνες. Ε, ωστόσο υπάρχει ακόμα δυνατότητα απάτης. για το θέμα της ανταλλογής εκπομπών. Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι ε, η, ακόμα και η ανταλλαγή εκπομπών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος. Ε, κάτι ακόμα το οποίο διαπιστώσαμε με αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά ε, ε, εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ότι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος και γίνεται με συστηματική απάτη και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει εκμετάλλευση και να υπάρξει απάτη και σε αυτές τις αγορές. Διαπιστώνουμε επίσης ότι ότι ακόμα και στους όρους ε, καταχώρησης ε, στα Μητρώα ε, μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο απέτης, γιατί σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει ένα Μητρό, αλλά υπάρχουν αρκετά και επομένω υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Υπάρχει και πρόβλημα με τις φορολογικές αρχές, διότι κάποιες φορολογικές αρχές σε κάποια κράτη-μέλη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να διαπιστώσουμε αν υπάρχει απάτη και να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ φορολογικών αρχών οι πληροφορίες αποτελούν στοιχείο κλειδί για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μορφή την απάτη. Επειδή στο συγκεκριμένο τομέα διακυβεύονται και πάρα πολλά χρήματα, οι ομάδε του οργανωμένου εγκλήματος ε, ε, κατάφεραν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο πλέον. διαπιστώσαμε ότι τα χρήματα τα οποία προέρχονται από αυτήν τη μορφή της απάτης τελικώς χάνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν δυνατότητα για, ε, εταιρείες για εταιρείε offshore, ε, χώρες στις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε γιατί δεν υπάρχουν ε, συμφωνίες διμερείς για συνεργασία και ακόμα και όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα χρήματα διαπιστώνουμε ότι έχουν φύγει σε χώρες με τις οποίες δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε εύκολα. και αυτό φυσικά δυσχεραίνει το έργο και των φορολογικών αρχών αλλά και των δικαστικών αρχών διότι εμείς απλώς προσπαθούμε να ρίξουμε λίγο φως σε αυτές τις υποθέσεις και δυσκολευόμαστε. Σε αυτή τη μορφή της απάτης λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια λύση σε εθνικό και μόνον επίπεδο. Προκειμένου να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Οι απαταιώνες δραστηριοποιούνται διεθνών και διεθνώς και επομένω ε, θα πρέπει να υπάρξει διεθνή συνεργασία και από πλευράς αρχών για να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα στην απάτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα συναλλαγών, μεταφοράς κονδυλίων, δεν υπάρχει πλέον κανένα σύνορο και από την άλλη, τα κράτη-μέλη και οι αρχές οι οποίες πρέπει να καταπολεμήσουν την απάτη πάντα έχουν σύνορα και όρους. Και όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία πράγματι δεν έχει φυσικά σύνορα εντός ε, ε, της επικράτειάς της, αλλά και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων των αρχών ε, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα, τα πράγματα που μπορεί να κάνουν οι αρχές σε διεθνές επίπεδο, διότι οι φραγμοί εξακολουθούν να υπάρχουν. Όπως είπαν και οι Βέλγοι συνάδελφοι, στη διοίκηση μπορέσαμε να προχωρήσουμε, μπορούσαμε να καθορίσουμε κανόνες ε, σε θέματα διοικητικής συνεργασίας από το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουμε το Eurofisc που γίνεται αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, μπορούμε να στείλουμε αιτήματα επαλήθευσης, μπορούμε να κάνουμε και κοινή επαλήθευση σε αρκετές χώρες, ε, μπορούμε να κάνουμε και ε, πολυμερείς παρεμβάσεις. Υπάρχει μια σειρά από κανόνες λοιπόν που μας λύνει λίγο τα χέρια. Ε, υπάρχουν αρκετές ε, δυνατότητες για να αγγιηθούμε τα εισοδήματα και να ε, διαθέτουμε και κάποια στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Από δικαστική σκοπιά τώρα υπάρχουν και συστήματα τα οποία μας επιτρέπουν να υπάρξει συνεργασία σε δικαστικό επίπεδο. Ε, υπάρχει επίσης η δυνατότητα δίμευσης, ε, συνεργασία σε θέματα ε, δίμευσεων. Και φυσικά υπάρχουν και η Europol και η Eurojust που μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι οργανισμοί. Όλα αυτά καλά, αλλά διαπιστώνουμε επίσης ότι οι εθνικές αρχές δεν αντιλαμβάνονται όλες απαραίτητα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ας δούμε για παράδειγμα τις φορολογικές αρχές σε κάποια κράτη-μέλη. Ορισμένε φορέ διεπιστώνουμε ότι έχουν μόνο διοικητικέ αρμοδιότητε και μπορούν να κάνουν μόνο φορολογικέ έρευνε. Δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα και να κάνουν και έρευνε τόπου, επί παραδείγματι, ή ε, κάποια ανάκριση. Ε, να δουν τι συμβαίνει σε ποινικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αστυνομία και φορολογικών αρχών. Ενώ σε κάποια άλλα κράτη-μέλη είναι διαφορετική η κατάσταση και εκεί οι φορολογικέ αρχέ έχουν και αστυνομικέ αρμοδιότητε σε κάποιου τομεί και μπορούν να κάνουν και έρευνε επιτόπου. Ε, αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην Ιταλία, στη Γερμανία. Στη Δανία όμω όχι. Και κατά συνέπεια, εάν υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, ε, υποθέσεις οι οποίες είναι αρμοδιότητα δύο χωρών, ε, π.χ. της Γερμανίας και της Δανίας, είναι δύσκολο να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών, διότι δεν υπάρχουν οι ίδιες αρμοδιότητες σε επίπεδο διοίκησης. Αν είναι η κοινέ οι αρμοδιότητε σε διοικητικό επίπεδο, τότε μπορούν να συνεργαστούν. Αλλά ε, μεταξύ Γερμανία και Δανία είναι αδύνατο, διότι η Γερμανία έχει περισσότερε αρμοδιότητε για τι φορολογικέ του αρχέ, ενώ εμεί όχι. Και αυτό είναι πρακτικό πρόβλημα. Ε, το ξέρω ότι έχω αντλήσει το χρόνο που μου δίνετε, αλλά ήθελα να σα δώσω και ένα παράδειγμα για να σα εξηγήσω τι εννοώ. Α πάρουμε για παράδειγμα τη Europol. Ε, υπάρχει μια ομάδα που κάνει αναλύσεις και ασχολείται με την κυκλική απάτη ΦΠΑ. Οι φορολογικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες. Εγώ συμμετέχω, πολύ ωραία όλα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε μόνο με καθοστό παρατηρητή. Και γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση που να επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να ανταλλάσσει πληροφορίες με τη Europol. Δεν υπάρχει επίσης και νομική βάση που να μας επιτρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες στα πλαίσια της συνεργασίας του Eurofisk με τη Europol ή το αντίστροφο. Και είναι λυπηρό αυτό, διότι δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της απάτης. Ε, με τα όργανα που έχουν στη διάθεσή μας στη σήμερα ημέρα, θα μπορούσαμε ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε μεγαλύτερο επίπεδο εναρμόνισης της νομοθεσίας και επίσης να εναρμονίσουμε τις αρμοδιότητες των διαφόρων αρχών γεγονός που θα μας επιτρέψει να έχουμε πραγματικά διασυνοριακή συνεργασία σε οριζόντιο επίπεδο ε, για την καταπολέμηση της απάτης. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίλσεν και τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας, ο κύριος Τόμας Γκάιερ. Μια στιγμούλα για να ανοίξουμε πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να μιλήσω στους ε, κυρίους και κυρίες βουλευτές. Πρέπει να πω για τους τρεις πολελαϊσάντες πως είναι πασίγνωστοι στην Ευρώπη και πολύ εξειδικευμένοι στον τομέα τους και είναι δύσκολο να προσθέσω εγώ κάτι. Οπότε θα περιουστώ σε ένα μικρό πραγματάκι. Δεν θα αφαιρθώ στα προβλήματα της φορολογικής διοίκησης, αλλά μόνο στα προβλήματα της ποινική δίωξης και ειδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας εισαγγελέα. Και αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα είναι 45 χρόνια διαφορά. Αυτό ήταν ο πρώτος φορολογικός κώδικας που μου έδωσαν εν έτη 1967 στο πρώτο εξάμεινο και αυτό εδώ πέρα είναι η του 2012. Βλέπετε λοιπόν πως ασχολούμε 45 χρόνια με την νομοθεσία, την φορολογική και τα της φοροδιαφυγής. Όταν με προσκάλεσαν σκέφτηκα πως να ξεκινήσω και σκέφτηκα τρία πράγματα. Υπάρχουν μια ταινία ε, στην οποία βοήθησα πριν από 10 χρόνια όταν γυρίστηκε στο σενάριο και ε, πήρε τρία χρόνια από την ζωή μου η υπόψη αυτή όχι η ταινία ήταν το μεγαλύτερο τότε φορολογικό καρουσέλ στην Ευρώπη είχαμε τότε στη Γερμανία. Βλέπετε εδώ πέρα την ταινία, βλέπετε τρία πλάνα από την ταινία. Κοιτάξτε το δεύτερο δεξιά. Ε, βλέπετε πως έπαιζε ο Φράνκο Νέρο. Αυτός είναι ο Φράνκο Νέρο, όταν ήταν ακόμα νέος και ωραίος, όπως ήμουν και εγώ τότε. Και περνάμε στον ε, υποψήφιο του S5 για την καγκελαρία στην Γερμανία, ο οποίος πριν από 15 μέρες ε, μίλησε στην τηλεόραση πάλι για το θέμα της απάτης του ΦΠΑ και τρίτον το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρθηκε πριν από μια εβδομάδα στις ε, εφημερίδες, στην εφημερίδα Handelsblatt συγκεκριμένα και έγιναν εκεί πέρα εκτιμήσεις συγκεκριμένες για το ύψος της απάτης ε, στον φόρο κύκλου εργασιών, όπως ε, λέγαμε τον ΦΠΑ. Και άρχισε το ελεγκτικό συνέδριο να ασχολείται με την αλλαγή της νομοθεσίας στις αρχές του 1994 και αυτό λόγω του ύψους της ε, απάτης. Και ε, όπως σας ανέφερα η υπόθεση που με απασχόλησε και έγινε ταινία ε, πήρε πολλά χρόνια από την ζωή μου σε μία ημέρα μάλιστα κάναμε έφοδο σε 224 γραφεία με 1500 αστυνομικούς στην Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και την Γερμανία. Και αυτό εδώ πέρα το σκαρίφημα ήταν οι σχέσεις και οι οικονομικές ροές τριών μηνών μόνο της απάτης αυτής. Βλέπετε πώς είναι το σχεδιάγραμμα. Και στο καρουσέλ αυτό είχαμε γύρω στα 40 εκατομμύρια τα οποία ανακτήθηκαν τότε. Και εκεί πέρα ξεκινούν τα προβλήματα. Κοιτάξτε, έχουμε τους απαταιώνες οι οποίοι μιλάνε πρώτα απ' όλα πολλές γλώσσες. Είναι σε πολλές χώρες. Σε μία δίκη μόνο είχαμε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Πρέπει να το... Ε, έχουμε το πρώτο πρόβλημα δηλαδή, αυτό τη συνεννόηση και αυτό το οποίο κάνω εγώ σήμερα, κάνω τρία πράγματα. Βοηθάω το Υπουργείο Οικονομικών, ασκώ διώξεις και προσπαθώ να ανακτήσουμε χρήματα. Και καταφέραμε να φέρουμε πολλά εκατομμύρια, να ανακτήσουμε πολλά εκατομμύρια από την Ελβετία, που είναι ιδιαίτερος δύσκολο να πάρει κανείς λεφτά που είναι κατατεθειμένα στην Ελβετία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ξεκινάμε από το προσωπικό. Δηλαδή, ο εισαγγελέα έχει διαφορετική εκπαίδευση από τον υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών και πάλι αυτοί οι δύο κάτι διαφορετικό από τον αστυνομικό. Αυτές οι τρεις αρχές επίσης έχουν διαφορετικές δομές διοικητικές εσωτερικά. Μετά έχουμε την ιδιαιτερότητα. Ο απλός εισαγγελέα δεν έχει φορολογικές γνώσεις, ούτε και ο αστυνομικό. Και σας είπα σας τα ξανάδειξα, εγώ ασχολούμαι 45 χρόνια με το φορολογικό δίκαιο και θεωρώ πως ε, είμαι από τους λίγους στην Ευρώπη εισαγγελείς που τέτοια εμπειρία. Και αντιστρόφως, το Υπουργείο Οικονομικών και οι εφορίες δεν έχουν νομικές γνώσεις. Τα επόμενα προβλήματα μετά στη δουλειά μας είναι ο μέσος εισαγγελέα αστυνομικός και εφοριακός, έχει κάποιες μέτριες γνώσεις αγγλικής. Δεν ξέρει ούτε Ολλανδικά, ούτε ξέρει να εκφραστεί στα γαλλικά. Τα ισπανικά του είναι κάτι το τελείως ξένο, να μην μιλήσουμε καν για τα πορτογαλικά. Και μετά έχουμε το επόμενο ζήτημα. Εγώ δεν ξέρω την ξένη νομοθεσία κατά κανόνα, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και οι φορολογικές αρχές και οι εισαγγελικέ αρχές έχουν τώρα το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο κανείς δεν δουλεύει πάνω στο ίδιο αντικείμενο πάνω από πέντε χρόνια. Τι σημαίνει αυτό. Μεγάλη εναλλαγή του προσωπικού. Δηλαδή, ο μέσος εισαγγελέας ξέρει λίγο απ' όλα και τίποτα δεν το ξέρει καλά να το κάνει. Και έχουμε άρα ουσιαστικό θεωρητικό οπλισμό αλλά και πρακτική πείρα ε, ελάχιστη. Ε, κοιτάξτε, εγώ σας είπα για την υπόθεση αυτή γεμίσαμε κοντέινερ με φακέλους και μετά είχαμε και αυτά που μας έστειλαν οι άλλες αρχές από άλλες χώρες. και στέλνει μετά το Υπουργείο Οικονομικών τους δικούς του υπαλλήλους στην Γερμανία ή στην Βρυξέλλες ή δεν τους το επιτρέπει. Οπότε τι κάνουμε. Ζητάμε μετά νομική αρρωγή από τους συναδέλφους μας. Αν μου επιτρέπετε να κρίνω λίγο το σύστημα αυτό της νομικής αρρωγής, έτσι, θεωρητικά θα έλεγα α, πως η κατάσταση είναι γενικά ικανοποιητική. Αλλά άνα χώρα, άνα περίπτωση, η κατάσταση κυμαίνεται από πάρα πολύ καλή μέχρι ελλειπής. Και δεν θέλω τώρα να αναφέρω συγκεκριμένες χώρες, γιατί δεν μπορεί η δικιά μου εμπειρία να είναι αντιπροσωπευτική. Αν με ρωτήσετε βεβαίως να σας πω να επενέσω κάποιες, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, η συνεργασία με την Ιταλία είναι υποδειγματική συνολικά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε επίσης είναι πως οι διαδικασίες ε, της νομικής ε, αρρωγής είναι μακροσκελής. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο και μετά υπάρχουν μεμονωμένες δυσκολίες. Ε, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις που δεν είναι ίδιες και στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο στο φορολογικό δίκαιο, μετά υπάρχει διαφορετική δικονομία, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και τα λοιπά διαφέρουν και μετά έχουμε, ή εγώ έχω εν πάση περιπτώσει, μεγάλα προβλήματα με το ζήτημα της ανάκτησης των χρημάτων. Θα σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα η Ελβετία μου δίνει τα λεφτά πίσω μόνο εάν υπάρχει απόφαση ποινικού δικαστηρίου και όχι φορολογικού. Δεν τους επαρκεί. Η Ολλανδία δεν μας βοηθάει στην ανάκτηση χρημάτων. Λένε, εγώ θέλω να μιλήσω με το Υπουργείο Οικονομικών. Και φαντάζεστε, με 26 χώρες τι διαφορές υπάρχουν στην νομοθεσία το οποίο τελικά καταλήγει να λειτουργεί προς όφελος του απατεώνα και εις βάρος των διοκτικών αρχών. Και αφού αναφέρθηκα σύντομα στα προβλήματα θα ήθελα 2-3 λεπτά να με ακούσετε για να προτείνω πιθανώς λύσεις. Η απλούστερη λύση είναι η Εγώ θα ήθελα σε ολόκληρη την Ευρώπη να υπάρχει ένα μητρό για τα ονόματα εταιριών και προσώπων. Κάτι ανάλογο με το σύστημα Eucaris. Το European Car Information System δηλαδή, όπου οποιαδήποτε χώρα είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, πατάει ένα κουμπάκι και διαπιστώνει ποιο αμάξι με ποιο, ποιον αριθμό πλαισίου βρίσκεται σε ποια χώρα. Το ίδιο θα ήθελα να ξέρω και σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η απλούστερη λύση. Βεβαίω, έχω και το ιδανικό, το όνειρό μου ενιαίοι νόμοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Nach. Εγώ, μετά από 45 χρόνια, δεν θα το ζήσω, αλλά σας παρακαλώ εσάς να το κάνετε. Υπάρχουν πρώτες προσπάθειες ήδη. Αναφέρθηκε το πρόγραμμα Φισκάλης. Ε, είναι η πανευρωπαϊκή συνεργασία η οποία έχει ήδη υπάρξει. Το δεύτερο είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Αλλά και εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα. Το τρίτο έχουμε τη συμφωνία του Στρασβούργου της 16ης Απριλίου, 16 Απριλίου και εκεί πέρα υπάρχει η δυνατότητα, αν διαβάσετε το άρθρο 10 τα έχω βάλει σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά όπου λέει πως επιτρέπεται ο εισαγγελέα ή εφοριακές αρχές χωρίς πρώτερη υπηρεσιακή βοήθεια ή νομική αροχή να ε, μάθει αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται αυτό σε ορισμένες χώρες. Δηλαδή, τι κάνω εγώ ορισμένες φορές. Στέλνω πληροφορίες ή παίρνω τηλέφωνο στην ξένη αρχή και λέω στείλτε μου ένα αίτημα για να σας δώσω πληροφορίες που μπορείτε εσείς μετά να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει επίσης και η Σουηδική πρωτοβουλία, η οποία θα είναι επιτυχής αν εφαρμοστεί και αυτό το οποίο θα ήθελα είναι μια ευρωπαϊκή αρχή. Αρμόδια. Μπορούμε βεβαίω ε, το να συζητήσουμε το αν θα είναι μόνο φορολογική αρχή ή αυτό το οποίο εγώ θα προτιμούσα μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όχι επειδή εγώ θέλω να γίνω Ευρωπαίος Εισαγγελέας, αλλά γιατί κατά την απόψή μου είναι η μοναδική δυνατότητα να γινω ευρωπαιος εισαγγελεα αλλα γιατι κατα την αποψη μου ειναι η μοναδικη δυνατοτητα να κυνηγησουμε τους δράστες εγκαίρως και μεταξύ της απλής και της ιδεώδους λύσης υπάρχει ενδιάμεση. Δηλαδή,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 αγαπητέ κύριε. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση μέχρι να φτάσουμε στην ιδέα όπως είπα. Να βοηθάει ο Όλαφ. Και θα εξηγήσω γιατί. Από όσο ξέρω, τότε, στον Όλαφ, είχαμε τους λεγόμενους δικαστικούς. Εισαγγελείς ή ε, ε, δικαστές εισαγγελείς που μιλούσαν πρώτον από κάθε χώρα μιλούσαν πρώτον την γλώσσα τους και δεύτερον ήξεραν σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ στη χώρα τους και βεβαίως ήξεραν και την εθνική τους νομοθεσία. Οπότε, όσο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ζητάω το εξής. Ενισχύστε τον Όλαφ, δώστε του τις εξουσίες έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει κάθε εισαγγελία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστούμε κύριε Σαγγελέα. Να ξεκινήσει η συζήτηση. Ποιο θέλει το λόγο, η κυρία Βάιλερ. Um Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη γιατί πρέπει να πάω σε άλλη συνεδρίαση, αλλά ο συνάδελφος εδώ, ο κύριος Βάιτεν Χόλτζερ, θα μου μεταφέρει την απάντησή σας. Άκουσα προσεκτικά τους ειδικούς και έχω δύο ερωτήσει προ τον Γερμανό, ε, τον κύριο Σεγγελέα, τον Γερμανό εμπειρογνώμονα. Κοιτάξτε, φοβήθηκα όταν άκουσα από εσάς πως ε, το Υπουργείο Οικονομικών τη Γερμανία. δεν επιτρέπει στους ε, εφοριακούς να μεταβούν στις Βρυξέλλες. Αυτό πρέπει να μου το εξηγήσετε. Ναι, αυτή, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, εγώ προέρχομαι, κατάγομαι από το κρατήδιο της ΕΣΥΣ. Ναι, το, το ξέρω τον Υπουργό Οικονομικών μας. Ναι, θα, θα τις κάνω όλες μαζί τις ερωτήσεις. Η εμπειρία που είχατε εσείς ε, με τον Όλαφ είναι και η δική μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι υπάρχει και θέλουμε να τον επεκτείνουμε. Γνωρίζετε επίσης πως ε, προγραμματίζουμε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ε, Προβλέπετε αυτό ήδη στη συνθήκη του Λουξεμβούργου, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς που ασχολείστε καθημερινά με αυτά τα ζητήματα. Τι θα έπρεπε μετά να έχει μια τέτοια αρχή ως αρμοδιότητες, ε, ως ε, διατάξεις, γιατί ένα όνομα μόνο δεν φτάνει. Δεν με ακούτε? Ε, τι ουσία δηλαδή θα έχει η αρχή αυτή. Αυτό θα ήθελα να γνωρίζω. Και μετά είπατε πως ε, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες ε, είναι δύσκολο να συνοηθούν οι ειδικοί γιατί οι μεν ξέρουν μία πτυχή και οι δε μία άλλη. Αλλά μα νομίζω πως για κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μία λεγόμενη task force, μία ομάδα δράσης δεν ξέρω ίσως να έχω ψευδεστήσεις για το τι μπορεί να επιτύχει, αλλά νομίζω πως υπάρχουν ειδικά για περιπτώσεις ε, φορολογικής απάτης ε, ή την απάτη με το διοξίδιο του άνθρακα κτλ. Το διάβασα αυτό, πως υπήρχε μια ομάδα δράσης που είχε και εφοριακούς και αστυνομικούς και εισαγγελείς μαζί για να ε, σχηματίσουν μια ομάδα τέτοια. Πείτε μας λοιπόν τι λείπει, ποιες είναι οι ελλείψεις και τέλος απευθυνθώ στους ε, άλλους ε, κυρίους. Νομίζω ο κύριος από την Ολλανδία είπε πως πρέπει να ε, χτυπήσουμε το φαινόμενο στη ρίζα του. Και βεβαίως αυτό δεν είναι μόνο η διασυνοριακή συνεργασία, αλλά σημαίνει και διαφορετικούς νόμους. Δηλαδή, έχουμε, από ό,τι φαίνεται, τελείως λάθος νομοθεσία για τον ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν έχουμε τόσο πολλές απάτες, σημαίνει πως και ο νόμος είναι λάθος. Και πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος το λόγο? Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ασχοληθεί με θέματα ΦΠΑ που είναι πολύ δύσκολο θέμα στην Ευρώπη γιατί έχουμε διαφορετικά συστήματα. Υπάρχουν κοινοί κανόνες αλλά διαφορετικά συστήματα σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και αυτό το καρουσέλ χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται τις διαφορές. Προσπαθούμε βέβαια να εφαρμόσουμε κοινού κανόνες για την καταπολέμηση του κλίματος και τα λοιπά, αλλά και των απατών, αλλά δεν νομίζετε ότι το αντίθετο θα έπρεπε να κάνουμε. Το όλο σύστημα του ΦΠΑ δηλαδή να αλλάξουμε. Γιατί τώρα προσπαθούμε να μπαλώσουμε απλώς. Στη χώρα μου από το 61 αν δεν απατώμε, οι Υπουργοί Οικονομικών είχαν πει ότι παρά το ότι περιοριζόταν στο 2% το σύστημα είναι πολύπλοκο και τώρα καταλήγουμε σχεδόν στο 25%. Μήπως θα έπρεπε να επιβληθεί μία ενωσιακή, ένας ενωσιακός ΦΠΑ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσουν όλα αυτά χωρίς να αντιμετωπίσουμε το καρουσέλ, χωρίς να αλλάξουμε το όλο σύστημα. Ο κύριος Φίλιψεν τώρα. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, ερώτηση της ε, Γερμανίδας ε, βουλευτού. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια ιστορία με μεγάλη... Πρόκειται για μια υπόθεση με μεγάλη ιστορία. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές ε, οδηγίες οι οποίες προσαρμόζονται συνεχώς, ειδικά οι εφαρμοστικές διατάξεις, ε, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από όλα τα κρατη Αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ είναι πως υπάρχει συχνά τελείως διαφορετική εφαρμογή από το ένα κράτος στο άλλο. Τώρα, ο Σπάλος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ε, προσπαθώ να δώσω κάποιες συμβουλές αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια παράδοση στα ζητήματα αυτά οπότε τι γίνεται ε, περνάνε προσωρινά μέτρα τα οποία κάνουν συχνά και ε, ευκολότερη την ζωή των απαταιών. Και συχνά επίσης ακολουθείται και η οδός της ίσονος ε, προσπάθειας και όσον αφορά την οργάνωση της διοίκησης και όσον αφορά την νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη, να σας πω τι είναι, ε, τι δίνει ε, αντικείμενο σε αυτή την απάτη είναι διαφορετικό το ποσοστό του ΦΠΑ που επιβάλλεται. Τα παιδικά τα ρούχα στο Ρωμανό Βασίλειο έχουν 0% ΦΠΑ. στι διπλανέ σκανδιναβικέ χώρες είναι διψήφιο. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα εύκολο ε, κίνητρο για εγκληματικές οργανώσει να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχουν εδώ πέρα αναρρύθμιτες δυνατότητες για απάτη. Για το δεύτερο ερώτημά σας, θα πρέπει να σκεφτούμε την μεταρρύθμιση του ε, συστήματος του ΦΠΑ. Ε, αν ε, μου επιτρέπετε, με κάθε σεβασμό έχουμε ένα προσωρινό σύστημα το οποίο ξεκίνησε το 1993 και βεβαίως καλύτερο θα ήταν να έχουμε ένα οριστικό σύστημα το οποίο θα δημιουργεί και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο θα διευκολύνει ειδικά τις εταιρείε οι οποίες δρούν με τρόπο διεθνή και θα καθαστήσει πολύ ευκολότερη τη ζωή των διοκτικών αρχών. Και ως κάποιος που δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να ζήσω και να συνεισφέρω σε ένα τέτοιο ομοιόμορφο ΦΠΑ. Αλλά όπως σας είπα είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα και με την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μέλων. Σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Λοιπόν, για το ερώτημα. Στο Ευρωφίσκ ακολουθούμε τη διοικητική οδό και η έγκαιρη ταύτιση προβλημάτων υπάρχει. Γνωρίζουμε από πολύ νωρίς ότι υπάρχει απάτη, αλλά πώς θα τη σταματήσουμε μπροστά σε οργανωμένο έγκλημα είναι δύσκολο. Δεν, σταμα... δεν αντιμετωπίζεται το έγκλημα με χαρτιά. Θα έπρεπε να μιλήσουμε ίσως αυτή την περίπτωση για υπερεθνικές δικαστικές αρχές. Και επομένως δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου κύριο Γκαγέρ. Γκάγερ. μικρόφωνο, κύριε Βάιλερ. Κυρία Βάιλερ. Για το ζήτημα της παρέμβασης άλλων αρχών που δεν έχει σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Να ένα παράδειγμα. Στη Βόνη, όπου εργάζομαι, βρίσκεται συμπτωματικά η κεντρική φορολογική διοίκηση. Και οι άνθρωποι εκεί είναι υπάλληλοι του Ομοσπονδιακού κράτους. Οπότε πρέπει τα υπηρεσιακά τους ταξίδια στις Βρυξέλλες να τα εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ομοσπονδιακός. Και όταν κάποιος στο Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να πάνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου στις Βρυξέλλες, δεν επιτρέπεται. Και μένα μου το απαγορεύσει ο προϊστάμενός μου, δεν μπορώ να το κάνω, εκτός αν πάρω μια μέρα άδεια και έρθω εδώ πέρα με δικά μου έξοδα. Έτσι. Εάν τολμούσε κανείς να μου το αρνηθεί, γιατί δεν το έχει τολμήσει κανείς ακόμα. Συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα, έτσι. Ε, είναι λεπτομέρεια, αλλά μπορώ να σα δώσω πολλά παραδείγματα. Για παρέμβαση των εθνικών αρχών, ε, αλλά παρέμβαση άσχετη με την ουσία τη υπόθεση για να επανέλθω στο ε, ερώτημά σας όσον αφορά την Task Force τη λεγόμενη. Κοιτάξτε, εγώ και άλλοι, όχι μόνος μου, μαζί με 25 άλλους ανθρώπους, από την εισαγγελία, την εφορία και την αστυνομία, ήμασταν, συναποτελέσαμε μια τέτοια Task Force. Και είχα το όνειρο πως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πυρήνα στον οποίο θα έρχονταν νέοι συνάδελφοι, θα μάθαιναν τη δουλειά και θα μετέδαν τη γνώση. Όχι, αλλιώς γίναν τα πράγματα. Οι διαφορετικές υπηρεσίες κατέστρεψαν την δουλειά μας και για λόγους εγωιστικούς. Κάθε υπηρεσία δεν θέλει να μπαίνει άλλος στα χωράφια της όχι, η αρμοδιότητά μου είναι δική μου. Και αν έρθει ο εισαγγελέα Τόμα Γκάιερ, βρίσκεται σε μια ειδική μονάδα, μετά από τρει εβδομάδε ή τρει μήνε ή τρία χρόνια, θα αρχίσει να κάνει αυτό το οποίο θεωρεί αυτός σωστό. Όχι αυτό το οποίο θεωρεί σωστό σωστό ο προϊστάμενά του ή ο αρχηγό αστυνομία ή ο υπουργό οικονομικών. Τι κάνω όμω εγώ, εφαρμόζω αυτό εδώ πέρα το βλιαράκι, το φορολογικό κώδικα και αυτά τα οποία λέει η συνείδησή μου. Και, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία task force η οποία λειτουργεί στη Γερμανία, του συναδέλφου Γκόντερτ, στην Φραγκφούρτη, ειδικά για την υπόθεση των δικαιωμάτων εκπομπών. Αλλά, θα μου επιτρέψετε να κάνω, να φέρω την αντίρρηση ενός μικρού εισαγγελέα. Γιατί θέλει τόσο πολύ καιρό να ερευνήσουν και να ζητήσουν να δώσει λογαριασμό η Deutsche Bank, μέσα από την οποία κύλησαν τα λεφτά. Έχουν τσιμπήσει τους μικρούλιδες, καταδικάστηκαν αυτοί ήδη. Έτσι, αλλά συγγνώμη, ε, έτσι, αυτοί είναι οι στρατιώτες. Εγώ θέλω το στρατηγό. Και εδώ πέρα βλέπετε πως εντάξει, πάντα έχει κάτι για να παραπονιέται ο εισαγγελέα. Είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί ο εισαγγελέα. Τι θα ήθελα λοιπόν. Θα ήθελα όπως σας είπα να επιβάλλω μεγάλες ποινές κάθριξης και να μπορώ να ξαναπάρω τα λεφτά πίσω. Δεν είδα λοιπόν να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Δεν είδα να μαζέψουν τα λεφτά. Θα σας δώσω λοιπόν αυτό εδώ πέρα το δισκάκι και μπορείτε σε 90 λεπτά να δείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια διαδικασία αν μας επιτρέπετε βεβαίως να το κάνουμε. Αυτά για την ώρα. Έτσι, αν, αν απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσεν για να κάνει τη τελικά συμπεράσματα. Δεν θέλει να μιλήσει ο κύριος Νίλσεν. No. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο λοιπόν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Περιμένουμε τώρα να έρθει ο Επίτροπος Σεμέτα θα διακόψουμε για λίγα λεπτά ένα αναμονή του Επιτρόπου. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές.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 Riprendiamo la seduta. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Ήρθε ο Επίτροπος μέτα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τον τέταρτο γύρο τη συζήτηση κατά πολέμηση τη αταπάτης και τη φοροδιαφυγής και ε, η προστασία της, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος ΕΜΕΤΑ, Επίτροπος για Φορολογία και Τελωνιακή Ένωση και της ΟΛΑΦ ε, ε, θα μας ε, παρουσιάσει το θέμα αυτό. Έχετε μισή ώρα για την παρουσίασή σας και κατόπιν θα ξεκινήσει η συζήτηση. Thank you very much. Σας κατευχαριστώ, Πρόεδρε, και κύριοι βουλευτέ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας αυτή την ακρόαση. Η παρέμβασή μου σήμερα συνδέεται άρρηκτα με το θέμα που συζητούσατε. Γιατί θα μιλήσω για... I want to introduce... για τις απάτες στο ΦΠΑ που συνδέονται με το θέμα και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτές οι πρωτοβουλίες της Ένωσης βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στην καταπολέμηση οργανωμένου κλίματος, αλλά το οργανωμένο έγκλημα παίζει σημαντικό ρόλο στην απάτη. Και δυστυχώς η απάτη είναι κερδοφόρια δραστηριότητα. Η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο στην Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης χάνει 2.000 ευρώ κάθε χρόνο λόγω της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Γνωρίζοντα αυτά, η Κομισιόν ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο ένα συνοπτικό και φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που συνοδεύτηκε από δύο συστάσεις στα κράτη-μέλη. Πώς να αντιμετωπίσουν τους φορολογικούς παραδείσου και πώς να σχεδιάσουν τη φορολόγησή τους. Αυτό δίνει ένα σημαντικό μήνυμα στο ολόκληρο τον κόσμο ότι η Ένωση είναι παίρνει σοβαρά υπόψη της το θέμα της φοροδιαφυγής και δείχνει ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία σε διεθνή βήματα, ιδίω στον ΟΣΑ, για να καταπολεμηθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Περιγράφει πάνω από 30 μέτρα για να αυξηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφάνεια, να θεσπιστούν κανόνες συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι και ένα ενωσια... ένας ενωσιακός αριθμός φορολογικής ταύτισης ή ταυτότητας. Επίσης προτείνει περισσότερη διαφάνεια και πέρα από την Ένωση, πράγμα που θα βοηθούσε την αποφυγή της φοροδιαφυγής που εκμεταλλεύονται άλλα φορολογικά συστήματα λιγότερο διαφανή. Η επιτυχία των μέτρων αυτών θα καθοριστεί από το βαθμό που θα δεσμευτούν τα κράτη-μέλη. Μόνο αν όλα συνεργαστούν πλήρως μπορούν τα μέτρα αυτά να επιτύχουν τους στόχους τους και γι' αυτό είναι ουσιώδες τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε κανέναν αριθμό ως προς το τι ποσοστό του ενός αυτού τρισεκατομμυρίου πηγαίνει στις τσέπες του οργανωμένου εγκλήματο ή των οργανωμένων εγκληματιών. Γνωρίζουμε όμως ότι το οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται και στην φοροδιαφυγή. Το σχέδιο δράσης λοιπόν περιλαμβάνει συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και του ξεκλίματο βρωμίκου χρήματο. Το μέτρο αυτό επιμένει ότι χρειάζεται σε έναρότερη συνεργασία μεταξύ όλων των διοκτικών αρχών και ιδιαίτερα των αρχών που είναι υπεύθυνε για την καταπολέμηση της ξεπλήματο βρωμικού χρήματο. Η συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών είναι ουσιώδη για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αντιμετώπιση φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και άλλων εγκλημάτων σχετικών με τη φορολόγηση. Το Ευρωπό, η Ευρωπόλ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών, συμβάλλοντα στην ταύτιση και καταστροφή των ε, εγκληματικών δικτύων. Πέρα από αυτά η Κομισιόν σχεδιάζει να αναφέρει συγκεκριμένα τα φορολογικά εγκλήματα ως προδρόμους του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος βάσει και των ε, συστάσεων του 12 της Financial Action Task Force. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια μιας νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση της τρίτης οδηγίας κατά του ξεπλήματος δρομικού χρήματος που σε λίγο θα παρουσιάσει η Κομισιόν. Αυτή η πρωτοβουλία θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των δικαστικών και δημοσιονομικών τιούτων για να αντιμετωπιστούν σοβαρές παραβιάσεις του νόμου. Η συνεργασία θα μπορούσε να διευκολυνθεί και περαιτέρω και από μια πανενωσιακή εναρμόνιση του αδικήματος του ξεπλήματος χρήματος με ανάλογες κυρώσεις. Και γι' αυτό η Κομισιόν θα προτείνει σύντομα μετά από την αθεώρηση της τρίτης οδηγίας αντιξεπλήματος χρήματος μια ειδικότερη οδηγία για την καταπολέμηση της το 2013. Άλλη δράση θα συνίσταται στον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών και λειτουργικής μεθοδολογίας για την ταύτιση των ροών χρημάτων από τις φορολογικές υπηρεσίες αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ταύτισης της χρήσης των πιστοτικών καρτών και των υπερακτίων λογαριασμών. Αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να διευκολύνει την ταύτιση των προβλημάτων, λαμβάνοντα υπόψη και την εμπειρία ορισμένων χωρών μελών για το θέμα αυτό, όπου υπάρχουν ειδικέ μονάδες για την δημοσιονομική πληροφόρηση. Κυρίε και κύριοι, όπω είπα και πριν, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της φορολογικής απάτης. Ε, Ανώ τις απάτες στο ΦΠΑ. Είναι βέβαια δύσκολο να υπολογίσουμε την επίπτωση αυτών των απατών, αλλά σύμφωνα με τους πρόχειρους υπολογισμού μας, το χάσμα, το έλλειμμα του ΦΠΑ μπορεί να αποτελεί μέχρι και το 12% του θεωρητικού ΦΠΑ που θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή περίπου 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το έλλειμμα είναι η διαφορά μεταξύ του θεωρητικού εσόδου από το ΦΠΑ για όλη την οικονομία και του πραγματικού εσόδου. Και μεγάλο τμήμα του ελλείμματος αυτού αφορά το καρουσέλ. Στο καρουσέλ οι επιχειρήσεις που θα έπρεπε να πληρώνουν το ΦΠΑ δεν το πράττουν. Και αυτό επιτρέπει σε άλλες εταιρείε στον αλυσίδα αυτή να εποφελούνται από χαμηλότερες τιμές. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε ότι η απάτη αυτή με τη μέθοδο του καρουσέλ απαιτεί συγκεκριμένες οργανώσεις, οργάνωση με πολλούς παράγοντες. Η επίπτωση είναι ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων στα κράτη-μέλη αυξάνεται και στρεβλώνεται και ο ανταγωνισμός στην αγορά. Το 2006 και 2008 η Κομισιόν πρότεινε μια ολόκληρη σειρά αντιαπατικών μέτρων για να καταστήσει πιο δύσκολο στους απατεώνες να εφαρμόσουν τέτοια μέθοδο καρουσέλου. Και πολλά από αυτά τα μέτρα τα ενέκρινε το Συμβούλιο. Αποτελούνται κυρίως από ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία του Ευρωφόρ, Eurofisk. Το κύριο καθήκον του Eurofisk είναι να ταυτίζει του, τα ελλείμματα στην αλυσίδα ως προς την πληρωμή του ΦΠΑ και επιτυγχάνεται από πολυμερείς ανταλλαγές ε, πληροφοριών για την έγκαιρη ταύτιση των προβλημάτων μεταξύ των χωρών μελών και ρόλος της Επιτροπής είναι να προμηθεύει στο Eurofisk τεχνική και λογιστική υποστήριξη. Εκτός από αυτό, το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροαπάτης ε, αναφέρει και ορισμένους νέους τομείς βελτίωσης, που είναι περισσότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, αντιμετώπιση νέων μορφών απάτης ως το δυνατόν συντομότερα μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης και μελέτης του πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα συστήματα φορολογικών εσόδων. Για το πρώτο, η Κομισιόν πιστεύει ότι οι Ευρωπαϊκέ Συμφωνίε με τρίτες χώρε για συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την απάτη στο διεθνέ εμπόριο, ιδιαίτερα ω προ το ΙΤΑ εμπόριο. Δεύτερον, τον Ιούλιο του 2012 η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για έναν Quick Reaction Mechanism που θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη να αναλάβουν ταχεία δράση κατά νέων τύπων καρουσέλ απάτης. Αυτός ο τα, μηχανισμός ταχείας αντίδρασης θα καταπολεμά σχήματα σχήματα προ-απάτης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των παραδοσιακών ελέγχων. Έτσι θα χορηγηθούν, γι' αυτό θα χορηγηθούν εξαιρέσεις στα κράτη-μέλη μέχρι και για ένα μήνα και το πολύ για ένα χρόνο. Οι συζητήσει στο Συμβούλιο δυστυχώ δεν έχουν ακόμη καταλήξει. Και αυτό κυρίω διότι μερικέ χώρε μέλη φοβούνται ότι θα χάσουν κυριαρχία. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν θα συνεχίσει να βοηθάει την Προεδρία για να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμβιβασμό. Τέλος, η Κομισιόν επίσης βοηθάει τα, υποβοηθά τα κράτη-μέλη για την καλύτερη φορολογική τους διαχείριση και αποτελεσματικότερη χορηγώντας τους τεχνική βοήθεια ιδιαίτερα όσον αφορά την μόρφωση των φορολογουμένων. Οι απώλειες από το ΦΠΑ που ζημιώνουν τα κράτη-μέλη είναι τεράστιες, αλλά και ο κοινοτικό προϋπολογισμός βλάπτεται από τις αφάτες στο ΦΠΑ. Ας δούμε λοιπόν τώρα, ας δούμε λοιπόν τώρα το θέμα του πώς θα προστατέψουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προεπλογισμό που συνεχίζονται ακόμη δείχνουν ότι και στο μέλλον θα πρέπει να εργαστούμε με λιγότερους αντί με περισσότερους πόρου. Άρα θα υπάρχουν λιγότερα μέσα εφαρμογής των προγραμμάτων που είναι ζωτικά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για τη δημιουργία ανάπτυξη και θέσεων απασχόληση. Η κατάσταση αυτή μόνο σε ένα συμπέρασμα μπορεί να μας οδηγήσει. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους πόρους που διαθέτουμε. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο στο ελάχιστο να, τελειώ, να καταλήξουν αυτά τα χρήματα σε λάθος χέρια. The EU's financial... Και το κύριο εργαλείο μας για να προστατεύσουμε τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης είναι η Όλαφ. Παρ' όλα αυτά η δουλειά της Όλαφ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική παρά μόνο να αναλυθεί αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών. Γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να συλλάβουν και να τιμωρήσουν τους απατεώνες. Κάτι με, δεν κάνουμε πολλά πράγματα σε κανέναν από αυτούς τους τομείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζήτησα την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το πρώτο στοιχείο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Εννοώ τη μεταρρύθμιση της Όλαφ, όπου υπήρξε πολιτική συμφωνία πέρυσι το Δεκέμβριο. Ελπίζω αυτό να μπορέσει να επισημοποιηθεί ως το δυνατόν συντομότερα. Γιατί όλα χρειάζεται αυτή τη νέα νομική βάση λειτουργία της για να είναι πιο αποτελεσματική. Άλλα μακροπρόθεσμα δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή Επιστρέφουμε στο εθνικό επίπεδο μόλις έχει κλείσει την, μια υπόθεση η Όλαφ και κάνει τις συστάσεις, και κάνει συστάσεις της. Παίζει λοιπόν το ρόλο του παρατηρητού σε εθνικές δικαστικές υποθέσεις και στις περισσότερες χώρες μέλη δεν μπορεί καν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που έλεξε η Όλαφ. Αντίθετα, οι εθνικές δικαστικές αρχές στην καλύτερη περίπτωση κάνουν τη δουλειά που έχει ήδη κάνει η Όλαφ και στη χειρότερη δεν κάνουν απολύτως τίποτα διότι οι απάτες κατά του ενωσιακού προϋπολογισμού είναι δύσκολο πράγμα και χρειάζονται πολλοί πόροι για τη διαπεραίωσή τους γιατί είναι διεθνείς περιπτώσεις. Γι' αυτό οι εθνικοί δικαστέ και οι εισαγγελείς μας λένε ότι προτιμούν να μην τις θεωρούν προτεραιότητες αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτόν τον λόγο τέτοιες υποθέσεις συχνά μένουν άλυτες. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Γιατί δείχνει ότι στην καταπολέμηση των απατών που ζημιώνει τον, τα, τους ενωσιακούς πόρους ε, κυριαρχούν ακόμη, αν και δεν αρκούν, εθνικές έννοιες. Πράγμα που δεν επιτρέπει την καταπολέμηση δύσκολων περιπτώσεων που από τη φύση τους είναι ενωσιακές και όχι μόνο εθνικές. Η συνάδελφός μου, αντιπρόεδρος Ρέντινγκ και εγώ, θα υποβάλουμε λοιπόν στην Κομισιόν τον Ιούνιο μία πρόταση για τον καθορισμό ενός, της θέσης ενός Ευρωπαίου Εισαγγελέα που λέγεται ΙΠΠΟ. Το, ο Ευρωπαίος αυτός Εισαγγελέας ΙΠΠΟ θα κάνει τις έρευνες, τις διώξεις που, ε, που αφορούν τον ενωσιακό προβλησμό πιο για να μπορεί χωρίς τις δυσκολίες που έχει τώρα να συλλέγει στοιχεία από όλα τα χώρα μέλη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και τους, την αναγκαία τεχνογνωσία για να το κάνουμε. Θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό αν είναι σε θέση να λειτουργήσει με βάση ένα πλαίσιο εναρμονισμένου ποινικού, ποινικού δικαίου. Αλλά τέτοιο εναρμονισμένο πλαίσιο θα ήταν επίσης σημαντικό και για διαμεθοριακές επιχειρήσεις εθνικά. Τον Ιούλιο του 2012 η Κομισιόν για αυτόν τον λόγο ενέκρινε μία πρόταση οδηγίας για την προστασία των ε, δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Με την πρόταση αυτή θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στο επίπεδο προστασίας του ενωσιακού προβλησμού από χώρα σε χώρα. Αυτή τη στιγμή οι καταδίκες που υποβάλλονται από την Όλαφ ε, για υποθέσεις που υποβάλλει η Όλαφ στα κράτη-μέλη πηγαίνουν από το 19% μέχρι το 92% ανάλογα με το κράτος. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στους διαφορετικούς ορισμούς των αδικημάτων, χαμηλές κυρώσεις και πολύ μεγάλους χρονικούς περιορισμούς που επιβάλλονται για την εκπαιδεύση. Οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο άρχισαν τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε ακόμη ορίσει κανέναν εισηγητή. Ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και για αυτό το θέμα για να βελτιωθεί η προστασία των χρημάτων των, καταναλωτών ε, φορολογουμένων. Για να καταλήξω τώρα θα ήθελα να στραφώ προ ένα άλλο σχέδιο που δεν αφορά το προπολογισμό τη Ένωση, αλλά ένα άλλο κοινό ευρωπαϊκό αγαθό, δηλαδή το ευρώ. Οι στατιστικές της ΕΚΤ δείχνουν ότι οι απάτες κατά του ευρώ, τα πλαστά ευρώ δηλαδή, παραμένουν σταθερές και η Ευρωπόλ επιβεβαιώνει ότι το αδιαπράττουν το αδίκημα αυτό κυκλώματα οργανωμένων εγκλήματος με τα δίκτυα που διαθέτουν. Γι' αυτό η Κομισιόν θέλει να προτείνει σύντομα μία οδηγία για την μεγαλύτερη προστασία του ευρώ. Το σχέδιο αυτό οδηγία θα προβλέπει περισσό, πιο αποτελεσματικέ έρευνες, περισσότερες και μεγαλύτερες κυρώσει και στεναρότερη εποπτεία τη εφαρμογής τη στα κράτη-μέλη. Για να συνοψίσω. Και η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής και για να προστατευτούν τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και η συμβολή σας στην επίτευξη του στόχου αυτού, επίσημη ή ανεπίσημη, είναι ζωτική. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να καταπολεμήσει την απάτη αποτελεσματικά από μόνο του. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται διαφάνεια και μια, και μια αποτελεσματική και γρήγορη ροή πληροφόρηση μεταξύ τους. Ιδιαίτερα πρέπει να δεχτούν ότι η αντιμετώπιση της απάτης δεν είναι θέμα απώλειας κυριαρχίας. Αυτή τη στιγμή οι απαταιώνες εποφελούνται από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών των κρατών μελών και εποφελούνται επίσης από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται και στη δικαστική συνεργασία. Δε αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Είναι καιρός να δράσουμε πια. Η Κομισιόν έχει προτείνει πολλά εργαλεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες μέλη. Πρέπει τώρα εσείς να πάρετε ταχείες αποφάσεις για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Σας έκανα μία περίληψη των δραστηριοτήτων μας και με χαρά να απαντήσω σε τυχόν απορίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Λέβα έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, διότι υπάρχει σλοβένικη καμπίνα στην συνεδρίαση. Τα καλά νέα καταρχάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει συγητή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε απάντηση στο πρόγραμμα δράσης που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τομέα της καταπολέμησης απάτης. Οι υποφαινόμενοι. Η έκθεση είναι σχεδόν έτοιμη, θα σας την παρουσιάσω στις 18 Φεβρουαρίου. Έχουμε εργαστεί σκληρά και με ιδιαίτερη επιμονή επί του ζητήματος και κάναμε και συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά τα ζητήματα αυτά και γνωρίζω και πολύ καλά το πρόγραμμα δράσης σας. Προσβλέπω λοιπόν στην ε, επικοδομητική συνεργασία μαζί σας και χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική και μια σαφή διαδικασία. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, απάτη. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους υπολείπους βεβαίως και υποστηρίζω πλήρως τα όσα έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω η εκθεσή μου ακόμα πρέπει να συζητηθεί και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν αλλαγέ, αλλά ε, θα παρουσιάζει την προσωπική μου άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ένωσης και θεωρώ ότι η διεθνής επίδραση της ε, ε, φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ε, είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Ε, μελετάω το θέμα αυτό εδώ και μήνες και διαπιστώνω ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, ε, μας απομένουν ακόμα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους φορολογικούς παραδείσους. Μπορεί να μην είναι βέβαια η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλο μέρος για να γίνει αυτό, αλλά θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί ο ορισμός του φορολογικού παραδείσου. Είμαστε στα 2013. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο name and shame, να κατανομάζουμε λοιπόν όσους είναι ένα δίκο. Ε, ποιοι είναι η φορολογική παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις γειτονές χώρες. Θα πρέπει να ακουστούν κάποια ονόματα. Και εγώ στην έκθεσή μου θα το τολμήσω. Θα τους κατονομάσω. Θέλω να ξέρω ποιες χώρες είναι φορολογική παράδοση, θέλω να υπάρχει ένας σωστός, κατάλληλος ορισμός και πρέπει να πάμε πέραν των συστάσεων που μας έκανε ο ΣΑ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και βεβαίως η φορολογική παράδοση έχουν να κάνουν και με τις μαύρες λίστες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μαύρες λίστες για τους φορολογικούς παραδείσους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υπάρχουν εθνικοί κατάλογοι. Εγώ όμως θα ήθελα να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ακόμα θέμα το οποίο ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αφορά τη Γερμανία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ε, για την άδεια τράπεζας που δίνεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε διαφυγή. Ε, θεωρείτε ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση. Τι άποψη έχετε. Ευχαριστούμε την κυρία Κλέβα και τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Ιακολίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Σαμέτα, ο οποίος ε, μας παρουσίασε εντό λίγων λεπτών μία σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις ε, πολύ συγκεκριμένε που θα μπορούσαν να ε, μας αποδείξουν και την ποιότητά του ως Επίτροπος. Μας έδωσε εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία. Κάθε χρόνο ένας πολίτης καταβάλει 2.000 ευρώ λόγω φοροδιαφυγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσό και φτάνει στο 1 δις ε, ευρώ και ε, φτάνει σε ένα 12% ποσοστό το οποίο δίνεται στην παράνομη οικονομία ενώ κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν την ευημερία των πολιτών. Μας αναφέρατε επίσης ε, ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερο συντονισμό για τα διεθνή αδικήματα, τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επίσης το νέο ρόλο της Όλαφ. Το ερώτημά μου λοιπόν αφορά τα δύο αυτά όργανα. Η Όλαφ είναι ήδη ε, ενισχύει και θα κάνει και μία ε, αναθεώρηση και ε, αυτό ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ε, προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εσείς και η κυρία Ρέντινγκ είστε οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν ότι το γεγονό ότι υπερασπιζόμαστε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το θέμα τη καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και την, ε, ε, τα νέα καθήκοντα τη όλα, αυτή θα φέρει ε, και για την νέα ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την Όλαφ και για τη Eurojust, ε, για όλα αυτά τα διεθνή αδικήματα τα οποία χρήζουν δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας που θα βαφίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και σας συγχαίρω. Τα καταφέρατε. Πείσατε Financial Times αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι λοιπόν επιτυχίες στο μέλλον. Είναι ένα πολιτικό ναρκοπαίδιο αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω εγώ μάλλον είμαι από τους ανθρώπους που πληρώνουν τους περισσότερους φόρους εντός της αιθούσης και αυτό εδώ και 40 χρόνια. Και όσο καταλαβαίνω το θέμα είναι θέμα στάσης, νοοτροπίας. Αν όλοι προσπαθούν να κλέψουν και θεωρούν πως οι φόροι πάνε κάπου αλλού και δεν με ωφελούν, ε βεβαίως θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Οπότε αυτός ο τομέας είναι περίπλοκος και όπως σας είπα είναι θέμα νοοτροπίας. Ε, πρέπει να ξέρετε πως εάν ε, βγάζει κανείς μεγάλους μισθούς πρέπει να, να έχει και κάποια αποτελέσματα ανάλογα. Αν δεν συμβαίνει αυτό ε, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρω ονόματα, το ξέρουμε. Και και τώρα να κάνω μια σύσταση, μου επιτρέπετε. Η Κομισιόν δεν πρέπει να το δει λίγο ευρύτερα. Και, και το Συμβούλιο. Γιατί κάθε πρόταση εδώ πέρα, βεβαίως, εντάξει, είναι πολύτιμη, αλλά αν αρχίσουμε να συζητάμε τον προπολογισμό της Ένωσης, χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά. Τα κράτη-μέλη δεν μας δίνουν Ξέρουμε πως υπάρχει φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και κάποιες χώρες ε, τα πάνε χειρότερα από άλλες. αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά και πούμε πως αυτά είναι τα χρήματα τα οποία χάνονται, δεν θεωρείτε πως ε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κοινή γνώμη και να οργανώσετε ε, και κάτι, γιατί όλες αυτές οι σύνοδοι κορυφής εστιάζονται σε ένα μόνο ζήτημα. Πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα. Και οι φόροι. Ε, συμφωνώ. Είναι ε, πιο σημαντικοί πλέον. Και οι εταιρείε ε, και τα λοιπά πρέπει να κάνουν αυτά τα οποία υπόσχονται. Εξού και η έλλειψη εμπιστοσύνη. Τι λέω λοιπόν. Ε, ίσως πρέπει να το δούμε ευρύτερα το ζήτημα. Ε, πρέπει να προσέχουμε ε, όταν λέμε πως από εδώ και από εκεί υπάρχουν φορολογική παράδειση. Στη χώρα μου έχουμε διπλάσιους φόρους από την Ιρλανδία όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Είναι φορολογικός παράδεισος. Σε άλλες χώρες ε, στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη ο φόρος είναι 20% για όλους. Εμείς έχουμε υπερδιπλάσιο. Εγώ πρέπει να πω πως ε, προς αυτές τις χώρες πως είστε από μια χώρα που είναι φορολογικός παράδεισος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Διστάζω. Και τέλος μια ερώτηση επιτέλους. Πρέπει να προγραμματίζουμε επιθετικά. Τι, τι εννοείται όταν λέτε επιθετικός φορολογικός προγραμματισμός. Εμείς είχαμε κάποτε ένα νόμο που έλεγε δεν επιτρέπεται ο φορολογικός ε, προγραμματισμός. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η νομοθεσία βεβαίω. Αλλά μιλήσατε για επιθετική φορολογική, φορολογικό προγραμματισμό. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να είστε κάπως πιο συγκεκριμένα, να μα εξηγήσετε τι εννοείτε. Ευχαριστώ, Ταβάρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σας δώσω ένα δύο λεπτά να βάλετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τη διερμηνία. Δεν ήμουν παρόν σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασής σας. Αναφερθήκατε στην ε, φοροδιαφυγή, δώσατε κάποια στοιχεία, αναφερθήκατε σε ένα 3 ευρώ. Είναι αυτό το ποσό. Πρόκειται για μεγάλο ποσοστό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Υπάρχουν όμως στοιχεία φοροδιαφυγής ε, ή μάλλον ποια είναι η αναλυγία μεταξύ φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για να γνωρίζουμε λίγο τι ε, χάνουμε σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και να σας πω ότι θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή αφορά κεντρικά ζητήματα της αγοράς, αλλά και ε, πλήττει και τη δημοκρατία το νομικό σύστημα που διαχειρίζονται το φορολογικά θετήματα είναι πολύ περίπλοκο και θα μπορούσε κάποιος ε, να ξεφύγει από το σύστημα. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις που έχουν ομάδες νομικών που ε, ασχολούνται αποκλειστικά με το πώς θα απαφύγουν τη φορολόγηση, ενώ οι απλοί πολίτες φυσικά δεν έχουν τέτοια μέσα στη διάθεσή τους. Υπάρχει λοιπόν μια συμμετρία ε, και στις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Αυτή η ασυμμετρία όμως ε, δημιουργεί και μια ε, ασυμμετρία εξουσίας και έχει και πολιτικές συνέπειες. Επομένως, υπάρχει διαφθορά, αλλά υπάρχει και διάβρωση των δημοκρατικών αξιών. Και αυτό φυσικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι διαβρώνεται, όπως είπα, το δημοκρατικό σύστημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρόβληματα είναι αρκετά χειρότερα διότι είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει. Στόχο μα λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά να έχουμε ένα πλούστερο σύστημα. Τα σύνθετα συστήματα οδηγούν σε ασυμμετρία εξουσία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πιο απλό σύστημα. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν μια ταπεινή πρόταση. Αυτή τη στιγμή 20 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μου, οι οποίες είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο, επομένως επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση ενημέρωσης ε, του κοινού, αποφάσισαν να μεταφερθούν στη χώρα του φίλου μου, του Ντενίς Ντογιούγκ, στις κάτω χώρες, γιατί εκεί δεν υπάρχει ε, υποχρέωση ενημέρωσης ε, και μπορούν απλώς να έχουν ένα ταχυδρομικό κώδικα και να είναι μια ε, letterbox company όπως αποκαλείται. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει πάρα πολύ ε, συχνά με τεγκαθίστατη επιχειρήσεις σε άλλες χώρες που έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις και είναι απλούστερα τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις όμως αυτές θα πρέπει να υποχρεούνται να δίνουν τις πληροφορίες που πρέπει να δίνουν βάσει και της δικαιοδοσίας ε, που ζητά περισσότερες πληροφορίες. Γιατί για παράδειγμα στην Πορτογαλία πρέπει να δίνουν ε, ένα σωρό πληροφορίες με τεγκαθίστανται στην ε, Ολλανδία και δεν χρειάζεται να δείσουν καμία από αυτές τι πληροφορίες. Δεν υπάρχουν λοιπόν οι ίδιες υποχρεώσεις. Τα τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Αν μια, χώρα, ε, ε, ε, μια επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο σε μια χώρα, θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Και κάτι συγκεκριμένο τώρα. Για το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, ο κύριος Σμιτ έχει δίκιο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η φορολογική παράδοση, αλλά υπάρχουν και μία σειρά από δυνατότητες ε, φοροαπαλλαγών γιατί είναι διαφορετικά τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και εδώ και πάλι υπάρχει διαφορά στις πληροφορίες. Υπάρχει η περιβόητη υπόθεση του SWIFT ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε πολυάριθμα μηνύματα στις Ηνωμένε Πολιτείες και ε, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται διμερώς και αμοιβαία όχι μόνο για θέματα καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας αλλά και για σοβαρά ε, διεθνή εγκλήματα και αδικήματα. Επομένως ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καταλήλως την νομοθεσία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία. Γιατί λοιπόν να μην τα χρησιμοποιήσουμε για να παίρνουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες όταν υπάρχουν οικονομικά εγκλήματα διότι οι Αμερικάνοι φίλοι μας μας ζήτησαν πάρα πολλά και πρέπει και αυτοί να μας δώσουν κάτι σε αντάλλαγμα, να μας δώσουν πληροφορίες όσον αφορά τα σοβαρά εγκλήματα. Αυτή είναι μια πρόταση που σας κάνω ε, και όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και με αυτό ολοκληρώνω, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα τμήμα έρευνας για οικονομικά αδικήματα ε, που να συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Europol ή ε, κάποιο άλλο όργανο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να διαθέτουμε ένα τέτοιο ε, τμήμα. Ένα ανακριτικό τμήμα για όλα τα οικονομικά εγκλήματα ε, ενός κάποια, μιας κάποιας εμβέλειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος mm, senza... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χωρίς να επεκταθώ σε εισαγωγές, θα ήθελα να κάνω πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις στον ε, αξιότιμο καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστώ και για τη σαφήνειά του και για τις ε, καλές προτάσεις που έκανε στη διάρκεια της παρουσίασής του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις ε, και βάσει των όσων μας είπαν κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες με τους οποίους μιλήσαμε. Παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε ένας εμπειρογνώμονας που έχει ψηλά καθήκοντα στον ΟΗΕ και για πολλά χρόνια ήταν διευθυντή ε, του ε, έρευνας σε επίπεδο ΟΗΕ για την ε, διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. και ο ειδικό αυτός, αλλά και άλλες πηγές, ε, θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, ε, μας λένε ότι η διακίνηση αυτής της μορφής δεν θα μπορούσε να συμβαίνει εάν δεν υπήρχε καθοριστικός ρόλος κάποιων τομέων του τραπεζικού ε, διεθνούς κυκλώματο. Και εδώ φυσικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τα θέματα για τα οποία συζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να παρέμβουμε. Το δικό σας το παρατηρητήριο τι μπορεί να μας πει για το ζήτημα, σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι έρευνά σα και τι μέσα θα μπορούσαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε ή να βελτιώσουμε προς αυτό το σκοπό. Και λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις σας, ε, παρά το γεγονό ότι αρκετές από τις παρατηρήσεις ε, της φιλοσοφίας της πολιτικής του κυρίου Σμιντ με βρίσκουν σύμφωνο, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να αναρωτηθούμε τι ρόλο διαδραματίζει η φοροδιαφυγή στην οικονομία των τραπεζών, στο τραπεζικό σύστημα. Εγώ γνωρίζω αυτά που μου έχουν συμβεί εμένα προσωπικά, όπως και οποιοδήποτε άλλο πολίτη της χώρας μου. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι είμαι αρκετά δραστήριος ε, ε πελάτης των τραπεζών της πόλης μου, όταν ήμουν και βουλευτής και στις τράπεζες στη Ρώμη. Ε, ποτέ δεν μου έτυχε να δω κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Παραδείγματο χάρη μία έκτακτη επιθεώρηση του ΔΟΕ στην ε, τράπεζα. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει ο φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος ε, ε, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και για μια μικρή απόδειξη εκατοντα, μερικών εκατοντάδων ευρώ και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν το σύστημα ελέγχου της φοροδιαφυγής να μην είναι και τόσο ε, προσεκτικό στα θέματα της διαφυγής που έχουμε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε και ποιος είναι ο ρόλος ε, των φορολογικών παραδείσων και θα πρέπει να παρέμβουμε εδώ χωρίς να είμαστε και ε, πολύ ακραίοι στις θέσεις μας διότι είναι γνωστό ότι είχαμε και πολύ κραυγαλές υποθέσεις. Ε, στη χώρα μου για παράδειγμα ο πιο μεγάλος επιχειρηματίας ε, στην τελευταία πεντηκονταετία και μάλιστα αυτές τις μέρες θα τον τιμήσουμε για τα 10 χρόνια μετά ε, από το θάνατό του, έναν άνθρωπο τον οποίο σεβομαι ιδιαίτερα, ε, αλλά από εκεί και πέρα με τα διάφορα κληρονομικά ζητήματα που προέκυψαν με τους ε, κληρονόμους του, διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που έκανε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Πρόκειται για τον Τζάνι Ανιέλη. Και υπάρχουν και αυτά τα περιβόητα κινέζικα κουτιά, μέσω των οποίων... Ε, κρύφτηκε και μέχρι τώρα δεν είναι σαφές ε, ποια ακριβώς είναι η διοκτησία της μεγαλύτερης αυτοβιομηχανίας ε, της Ιταλίας. Και αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ε, λόγο ως που έχουν οι φορολογικές αρχές και τι ελέγχουν τα σώματα δίωξης οικονομικού εγκλήματος, γιατί ορισμένες φορές υπάρχουν ε, και υποκρύπτονται και περιουσιακά στοιχεία. Δεν συμβαίνει αυτό για τη Fiat, για παράδειγμα, προς Θεού, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κρυφά κρυμμένα στοιχεία τα οποία να σε πρόσωπα τα οποία ε, έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και είναι προϊόν εγκλήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο γιατί θεώρησα πως συνάδελφοι θα κάλυπταν όλα τα ζητήματα, αλλά κάποιες παρατηρήσεις των συναδέλφων με κάνουν ε, να... θέλω να αντιδράσω με κάποιες επρόσθετες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, κύριε Σμιτ, εγώ πληρώνω πάρα πολλούς φόρους. δεν χρειάζεται νομίζω να το πω. Ε, σε ένα προϊόν βέβαια το οποίο είναι το, το πιο φορολογικά συμφέρον, αλλά έχει δίκιο ο κύριος ε, Σμιτ ε, εδώ πέρα, πως ε, πράγματι είναι φυσικό ο κόσμος να προσπαθεί να αποφύγει τους, τους φόρους. Αλλά κοιτάξτε, ε, το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή όταν μια πορτογαλική επιχείρηση χρησιμοποιεί ας πούμε, τις πορτογαλικές υποδομές έχει την ηθική υποχρέωση να τις πληρώνει. Και υπάρχει και αυτή η ηθική ε, πτυχή και πρέπει και η δική μας η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη. Καλό είναι να συνεννοηθούμε όλοι πως ε, η φόρο αποφυγή και η αναζήτηση χαμηλότερων δυνατών φορολογικών συντελεστών δεν είναι κάτι το και πρέπει να προσπαθήσουμε το καταπολεμήσουμε. Αυτό γίνεται με τη διαφάνεια, δηλαδή οι επιχειρήσεις να μας πούν άνα χώρα τι τζίρο κάνουν και τι φόρο πληρώνουν και όχι όπως τώρα ή όπως κάνουν συχνά οι πολυεθνικές να δουλεύουν με ομιχλώδη νούμερα και επιτέλους η Κομισιόν θα πρέπει να καταλήξει και σε μια οδηγία περί λογιστικής και να κάνει μια σχετική πρόταση. Δεύτερον, αυτό το οποίο είπαν οι συναδελφοί, το τι είναι φορολογικός παράδεισος. Ήμουν παρόν σε συζήτηση με την Ολλανδική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ομπάμα και μας ε, κατηγόρησαν, ε, μας κατηγόρησε ο πρόεδρος Ομπάμα ότι είμαστε ε, φορολογικός παράδεισος ε, και του αντίτινε, αντίτινε η Ολλανδική κυβέρνηση πως δεν είμαστε εμείς. Ε, μπορείτε να δείτε τον ορισμό που δίνει η ε, αρμόδια σχετική υπηρεσία η οποία δεν μας συγκρίνει πραγματικά με Κατάρ και λοιπούς πραγματικούς φορολογικούς ε, παραδείσους. Και βεβαίω ε, μην ξεχνάμε πως όταν προσπαθήσαμε να δούμε το τι πληρώνουν διάφορες πολυεθνικές, πολύ γνωστές, κατέληξε η γνωστή οργάνωση Tax Justice στο ότι πληρώνουν ένα 2%. Δεν πληρώνουν φόρους δηλαδή στην Ευρώπη, ούτε στην Ολλανδία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε πουθενά. Αυτό είναι απαράδεκτο κύριε Επίτροπε. Οπότε πρέπει να καθορίσουμε σωστά τον φορολογικό παράδεισο, αλλά και για τα δικά μας τα κράτη-μέλη. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς κρίνετε τις Ολλανδικές πρακτικές. Ε, εγώ θα τολμούσα να πω πως ε, πιθανώς είναι φορολογικός παράδεισος η Ολλανδία. Αλλά πρέπει νομίζω να καθορίσουμε πως ε, αυτές οι πρακτικές δεν είναι σωστές, ειδικά για βιομηχανικές χώρες όπως η ε, Ολλανδία και πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και ένα συγκεκριμένο σύστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Βάιλερ. Ναι, ένα σύντομο ε, ερώτημα και να με συγχωρείτε. Όταν προέκυψε αυτό το σκάνδαλο σε όλα τα ΜΜΕ, πως μεγάλες αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω του να αλλάζουν ε, χώρες ε, και θηγατρικέ ε, πληρώνουν μόνο 2% φόρο όπως η Starbucks ε, και η Shell και πολλές μεγάλες εταιρείες προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στα γερμανικά μνημεία και στα βελγικά. Σκοπεύετε κύριε Επίτροπε να υποβάλλετε μια οδηγία για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Ωραία. Εγώ, ακούγοντας και τις παρεμβάσεις των συναδελφών, δεν θα ήθελα... να ξεκινήσει μια μάχη εδώ ποιος είναι πιο καλός φορολογικός παράδοσος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί νομίζω ότι κάθε χώρα έχει κάτι να κρύψει και θα έπρεπε να τρέπεται γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πάμε στα νησιά Κεϊμάν. Έχουμε το Βατικανό, το Λουξεμβούργο, το Σαν Μαρίνο, την Ελβετία. Δεν είναι και στην άλλη άκρη του κόσμου όλες αυτές τις περιοχές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ εκτίμησα τα όσα είπε ο Επίτροπος και πρέπει να πω ότι τέσσερα χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και πρώτη φορά ακούω ο Επίτροπο να λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα έτσι να τα αλλάξουμε. Τα εκτίμησα ιδιαίτερα λοιπόν όλα αυτά και, τα... και εκτίμησα και ιδιαίτερα το φιλόδοξο τρόπο ε, με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα. Τολμάει και λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα αλλάξουμε πορεία. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει οικονομική κρίση διαστάσεων που δεν μας δίνουν πραγματικά καμία πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει η κρίση. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε 140 δισεκατομμύρια ετησίω μόνο στην Ιταλία τη χώρα μου, αυτό είναι το κόστος της μαφίας. Μόνο στην Ιταλία. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Και αυτά τα ποσά είναι και υπεκτιμημένα. Η Επίτροπος ε, Βάλστρο μας είπε ότι 150 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μας είπατε και αυτά τα αστρονομικά ποσά για τις ε, προβλέψεις για την ε, φοροδιαφυγή. Ζητάμε λοιπόν από τους πολίτες να πληρώνουν τους φόρους τους. Και δει να τους πληρώνουν και με, με κόπο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν και εμείς αξιόπιστοι. Να επενθυμίσω ότι έγινε πέρσι, μάλλον δύο χρόνια πριν, ε, με το φορολογικό ζήτημα, ε, το φορολογικό σκάνδαλο ε, ενώπιον του οποίου σήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν τεράστιο το σκάνδαλο για τη χώρα μου. Δόθηκε αμνηστία και κατάφεραν οι ίδιοι ε, γνωστοί να βγάλουν έξω το ε, κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, ε, παράνομα κεφάλαια και τα ξαναέφερε στη χώρα, αλλά δεν ξαναγύρισαν στα χέρια των φορολογικομένων, επιστράφηκαν στους απατεώνες. Και εγώ λοιπόν, όπως και ο κύριος Μπορκέτσιο, αναρωτιέμαι, αυτή τη στιγμή που πραγματικά οι πολίτες μας πιέζονται. είναι δύσκολο να είμαστε μάρτυρες στην φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρήσεων, ακόμα και μεγάλων τραπεζών. Εχθές και σήμερα στην Ιταλία συζητήθηκε το σκάνδαλο των παραγόγων της Μοντε Πάσκης Σιένα και πρόκειται για μια κατάσταση πραγματικά είναι ανυπόφορη, διότι αυτά τα μεγάλα κυκλώματα αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες δεν πληρώνουν, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλουμε φορολογία στη μικροεπιχείρηση την οικογενειακή, είναι πολύ πιο εύκολο ε, να επιβάλλουμε φορολογία στο μικροέμπορο και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο σκότωσε την οικονομία στην Ευρώπη. Προσέξτε, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά... Αυτή τη στιγμή εμεί ε, αυξάνουμε το ΦΠΑ, ε, μειώνουμε την αγοραστική αξία ή και την απειλούμε την αγοραστική αξία για τους πολίτες και ε, φορολογούμε μισθούς, φορολογούμε το, ε, πάρα πολλά πράγματα και δεν ξεκινάει μια σοβαρή μάχη χωρίς όρια όπως είπατε κι εσείς απέναντι σε όλους όσους ε, κάνουν μεγάλες κλίμακας φοροδιαφυγή. Ελοχεύει ο κίνδυνος κατά την άποψή μου να μην είμαστε πλέον αξιόπιστοι. Ελπίζω λοιπόν και με τη βοήθειά σας και με τα όσα άκουσα από εσά κύριε Επίτροπε, να υπάρξει πραγματικά μία σκληρή μάχη κυρίως κατά όλων αυτών που ε, κάνουν μεγάλη κλίμακα φοροδιαφυγή, διότι έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό το κενό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε που πρέπει να πάμε να βρούμε χρήματα αν πραγματικά θέλουμε να ανακτήσουμε ε, το έλλειμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε που, ποιοι είναι αυτοί που τα διαθέτουν. Και κατά την άποψή μου, τα κράτη-μέλη, όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να πιστέψουν, πρέπει να επενδύσουν, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και τα κράτη-μέλη ότι αυτή είναι η κυριότερη υπεύθυνη αυτού του οικονομικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όταν συζητώνται αυτά τα θέματα υπάρχουν ε, φραγμοί και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, διότι αυτό ζη... Ε, ζημίωσε τον... ε, τον Ιταλικό λαό, εισήχθηκε αυτή η δυνατότητα φορολογικής αρμνηστίας και χρησιμοποιήθηκε και αυτό έπληξε ε, πραγματικά τη στιγμή στην οποία ήταν δύο οικονομικέ επιχειρήσει εν εξελίξη και ε, όλοι έβαζαν χέρι στην τσέπη των Ιταλών πολιτών ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχαν παράνομα κεφάλαια στο εξωτερικό τα οποία επέστρεψαν στην Ιταλία με ένα ελάχιστο τίμημα, πραγματικά ένα μικρό ποσό δόθηκε, γελίο, ε, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατάκλεψαν τους Ιταλούς πολίτες. Ελπίζω λοιπόν να λυθεί το ζήτημα και αυτό να μείνει μόνο μια άσχημη ανάμνηση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα, να αναστρέψουμε την πορεία μας όπως είπατε εσείς. Σας δίνω και πάλι το λόγο για να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Αν με επιτρέπετε θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, κυρία κυρία Κλέβα. Ξέρω πως είστε η συγκήτρια. Και βεβαίως ε, εγώ μίλησα για την ε, ε, οδηγία προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν τον Ιούλιο. Τώρα έχουμε Ιανουάριο και ακόμα βεβαίω δεν έχουμε εισηγητή από το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Τέσσερα να είναι άλλο το αντικείμενο αυτό. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα αυτά που ετέθησαν σήμερα. Πιο γενικά μιλώντας, νομίζω πρέπει να αντιληφθούμε πως ε, στον τομέα της καταπολέμησης φορολογικής ε, απάτης και της φοροδιαφυγής βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολλά στο επίπεδο της Ένωσης αλλά ε, χρειαζόμαστε και προσπάθειες και σοβαρές προσπάθειες στο επίπεδο των κρατών μελών και οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες ε, πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει καλά μέσα, θα έλεγα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα έχετε μάλλον δει πως έχουμε σοβαρά στοιχεία φορολογικής πολιτικής και μέσω των συστάσεων αναχώρα δίνουμε στοχευμένες συστάσεις ε, στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τα ε, ζητήματα φοροδιαφυγής και απάτης στο εθνικό επίπεδο. Αυτό έγινε ήδη στο πλαίσιο του δεύτερου ευρωπαϊκού εξαμήνου και θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο ε, και με τρόπο πιο στοχευμένο τις προσπάθειες στο τρίτο ευρωπαϊκό εξάμεινο που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, για να επιστρέψουμε στο ζήτημα των φορολογικών παραδείσων, πολύ μιλήσατε για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, δώσαμε έναν ξεκάθαρο ορισμό του φορολογικού παραδείσου στις συστάσεις μας και προχωράει παραπέρα από τον ορισμό του ΩΣΑ, γιατί ο ορισμός του ΩΣΑ συμπεριλαμβάνει μόνο διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών και αυτή τη στιγμή η μαύρη λίστα του ΩΣΑ είναι άδεια ενώ ο δικός μας ορισμός ε, συμπεριλαμβάνει πάρα, πολλά, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία δηλαδή δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό αποφυγή του, των βλαβερών φορολογικών πρακτικών με συγκεκριμένα κριτήρια. Όταν λέω κριτήρια, τι εννοώ. Τα εξηγούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πρότασή μας. Και βεβαίως, όπως είπα, πηγαίνουμε πέρα από την πρόταση του ΩΣΑ και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο διεθνές πλαίσιο και οι ορισμοί μας ε, γίνονται δεκτοί ως διεθνείς ορισμοί. Και βεβαίως εννοείται ότι ισχύουν εντός της Και βεβαίως αναφέρθηκε και η ανάγκη να κατονομάσουμε. Ε, η μαύρη λίστα αυτό ακριβώς είναι. Η σύσταση μάλιστα ζητά από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μαύρες λίστες επικρατιών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν φορολογική παράδειση σύμφωνα με τον ορισμό μας. Και νομίζω πως επίσης είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη πως ε, πρέπει να κάνουμε προτάσεις ε, εντό ε, του πλαισίου των συνθήκων. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό καμιά φορά, ακόμα και αν θέλουμε, δεν μπορούμε να προτείνουμε κάτι το οποίο πιθανώς παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για μαύρες λίστες, εφαρμογή, και τις ε, συστάσεις ε, για τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό προτείναμε στην ανακοίνωσή μας ε, την σύσταση μιας πλατφόρμας για την χρηστή φορολογική διοίκηση με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων και επίσης ε, τον συντονισμό ε, της εφαρμογής και με τον τρόπο αυτό θεωρούμε πως ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε συντονισμένους καταλόγους, λίστες φορολογικών παραδείσων. Οπότε δεν είναι μόνο συστάσεις, αλλά όπως είπα και κάποιες δομές διοίκησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ε, συστάσεων. Και βεβαίως, ο κύριος Όλε Σμιτ έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για τις επιθετικές φορολογικές πρακτικές, όπως είπαμε, και τις σχετικές συστάσεις. Και ρωτάει τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Υπάρχουν γενικές ρήτρες μη κατάχρησης ε, στα κράτη-μέλη, κατά οποίο σημαίνει πως ε, κάποιες ε, συναλλαγές γίνονται μόνο για λόγους φοροαποφυγής και θα μπορούσαν να αγνοηθούν όταν μιλάμε για τον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης κάποιων εταιριών. Τι μιλάμε δηλαδή για την τεχνητή μεταφορά κερδών από τη μία χώρα στην άλλη με στόχο να αποφευχθεί ή να μειωθεί ε, το φορολογικό βάρος. Οι δύο συστάσεις αυτές θα συμπληρωθούν και με συγκεκριμένες προτάσεις για τροποποίηση της, ε, των οδηγιών, των οδηγιών, των εταιρικών των λεγόμενων, ε, δηλαδή οδηγία περί συγχωνεύσεων, ε, περί δικαιωμάτων χρήσης κτλ. Και θα το δούμε αυτό το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι πως εάν εφαρμοστούν ε, σωστά αυτές οι συστάσεις μαζί με την αλλαγή των εταιρικών οδηγιών θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα γνωστά προβλήματα που περιγράφονται στα ΜΜΕ και αφορούν τις μεγάλες πολυεθνικές ε, τη Google, τα Starbucks και τα λοιπά. Βεβαίω ε, τα ονόματα αυτά προσελκύουν την προσοχή, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείε λιγότερο γνωστές ε, που κάνουν, ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές. Αλλά βεβαίως δεν είναι τόσο ελκυστικές από πλευράς ε, πρωτοσέλιδων. Γενικώ λοιπόν, μιλώντα, θα έλεγα πως τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια μετατόπιση όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και απάτης και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, μόλις ετέθη ενισχύ η νέα οδηγία για την ε, διοικητική συνεργασία από 1η του 2013 και η οδηγία διοικητική συνεργασίας προβλέπει πρώτα απ' όλα καταργεί τραπεζικό απόρριτο γιατί σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν ε, να μην απαντούν πλέον σε αιτήματα για παροχή ε, πληροφοριών για λόγους ε, τραπεζικού απορρίτου. Αυτή είναι η βασική συνέπεια και μετά προβλέπεται και μία διεύρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς από 1ης Πρώτου 2015 θα συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως ε, αμοιβέ ε, συντάξεις, ε, εισόδημα από ιδιοκτησία και διάφορα άλλα. Και κάποια στιγμή αργότερα πληροφορίες για μερίσματα και κεφαλαϊκές αποδόσεις ε, κτλ. Βλέπετε λοιπόν πως η γενικότερη αντιμετώπιση ανταλλαγής ε, πληροφοριών ε, διευρύνεται. Και θεωρώ πως με τις πρόσφατες εξελίξεις και στις ΕΠΑ με την εισαγωγή της νέας ε, νομοθεσίας, ε, ο λεγόμενος νόμος ε, φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών, μας οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα με τις ΙΠΑ για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και στο παγκόσμιο πλαίσιο. Ξεχνάμε πως η φάτκα σημαίνει και αμοιβαιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ε, κάθε χώρας ε, και των ε, ΙΠΑ. Εάν η χώρα υπογράψει το λεγόμενο υπόδειγμα 1 στη συμφωνία υποδείγματος 1 δηλαδή διακρατικές ανταλλαγές πληροφοριών ε, στην ίδια κατεύθυνση λοιπόν πηγαίνουμε με τις ΙΠΑ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα με την οδηγία περί αποτομίευσης και την επέκταση της εντολής για διαπραγμάτευση με την Ελβετία. Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν ε, την ε, συμφωνία αλλά ελπίζω πως ε, με τις νέες διεθνείς εξελίξεις μπορώ να κατονομάσω τα κράτη άμα θέλετε. Κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε να γνωρίζουμε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τα ονόματα των χωρών που μπλοκάρουν των δύο χωρών. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Το λέω παντού, όπου μιλάω. Οι δύο χώρες είναι το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, πήγα στην Αυστρία και διαπραγματεύτηκα με τους αυστριακούς ε, συναδέλφους το ζήτημα αυτό Οπότε θα δούμε. νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος ε, στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και νομίζω πως είναι και προς το συμφέρον ε, των ε, κρατών μελών ε, που έχουν προβλήματα ε, στα δημόσια οικονομικά τους να μπορούν να συλλέγουν φόρους τους φόρους που οφείλονται κατόπιν έχει δίκιο ο Όλε στην παρέμβασή του ε, όταν μιλάει για την ανάγκη του να δούμε το ζήτημα ευρύτερα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά εγώ κατάλαβα πως εννοείται πως ε, οι φορολογούμενοι πρέπει να θεωρούν πως τα χρήματά τους ξοδεύονται σωστά. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο βεβαίως ε, θα βελτιωθεί και η εθελοντική συμμόρφωση. Συμφωνώ πλήρως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στην τομέα της διαφάνειας στην δημιουργία δυνατοτήτων ε, για να αντιληφθούν οι φορολογούμενοι που ξοδεύονται τα χρήματά τους και εδώ είναι ο ρόλος των αρχών των κυβερνήσεων να επιδείξουν δηλαδή πως τα χρήματα αυτά δεν τα σπαταλάνε αλλά πως πάνε σε επενδύσεις, ε, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ποιοτικές υπηρεσίες. Ε, γνωρίζω πως η Σουηδία είναι πολύ καλή σε αυτό. Και παρά την υψηλή ε, φορολογία, το επίπεδο της φοροαποφυγής είναι πραγματικά χαμηλό. Και μάλλον αυτό είναι και παράδειγμα νομίζω μιας χώρας η οποία συνδυάζει υψηλό επίπεδο φορολογίας και χαμηλό επίπεδο φοροαποφυγής. Τέλος, αναφέρατε την Ολλανδία και το ότι πορτογαλικές εταιρείες μεταφέρουν την έδρα τους στην Ολλανδία για το χύψη λόγο. Πρέπει να είμαι σαφής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα μέσο ακριβώς για να καταπολεμηθούν οι βλαβερές ε, φορολογικές πρακτικές. Γι' αυτό θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φορολογική παράδεισοι γιατί κώδικα συμπεριφοράς ε, για την φορολογία των επιχειρήσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζουν ποιες είναι οι βλαβερές ε, φορολογικές πρακτικές. Και από το 1997 έχουν αναλυθεί πάνω από 400 τέτοιες πρακτικές και πάνω από 100 από αυτές αναγνωρίστηκαν ε, ως βλαβερές. Και κράτη-μερή άλλαξαν αυτές τις πρακτικές για να συμμορφωθούν με τον κώδικα. Αλλά νομίζω πως το πρόβλημα είναι πως δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν ε, χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο με τρόπο αποτελεσματικό. Οπότε αν κάποια χώρα έχει προβλήματα με άλλη χώρα, χώρα θα μπορούσε να πάει στην ε, αρμόδια ομάδα, τη ε, λεγόμενη ομάδα κώδικα συμπεριφοράς και η άλλη χώρα μετά πρέπει να αναλύσει τη συμπεριφορά της από τη σκοπιά του δίκαιου φορολογικού ανταγωνισμού. Και εάν η πρακτική οριστεί ως βλαβερή, τότε θα πρέπει να αλλάξει. Οπότε θεωρώ πως πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε αναπτύξει μαζί και προτείνουμε μάλιστα να επεκτείνουμε και τον κώδικα συμπεριφοράς ε, στην ε, φορολογία επιχειρήσεων για να συμπεριλάβουμε και τα πλούσια άτομα πέρα από τις επιχειρήσεις γιατί έχουμε το πρόβλημα πως ε, και τα πλούσια άτομα μπορούν να μετακινήσουν το εισόδημά τους ε, για να μειωθεί το φορολογικό βάρος. Οπότε Τώρα θα ήθελα να στραφώ ε, στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Το ερώτημα του κυρίου Ιακολίνο για το μελλοντικό υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εξολόγηση αντικτύπου πολλά πιθανά μοντέλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινώντας με ένα πλήρως κεντρικό μοντέλο μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή κεντρική ευρωπαϊκές διαδικασίες και μετά υπάρχουν και άλλα μοντέλα πιο αποκεντρωμένα δηλαδή με μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο κέντρο και στα κράτη-μέλη. Αναλύουμε λοιπόν τα διάφορα μοντέλα στο πλαίσιο της αξιολόγησης αντικτύπου και με βάση αυτό μετά θα επιλέξουμε το καλύτερο μοντέλο. όσον αφορά τη Eurojust. Βεβαίω, η Eurojust ε, θα αποτελέσει μέρο τη μεταρρύθμισης γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πω η συνθήκη λέει πως ε, μια ευρωπαϊκή εισαγγελία μπορεί να δημιουργηθεί από τη Eurojust. Αυτό σημαίνει πως ε, η μεταρρύθμιση θα επηρεάσει και τη Eurojust ε, και τον Όλαφ. Και όλα τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε ερευνητικές δραστηριότητες. Ε, αλλά βεβαίως ε, πέρα μιλάμε και για ποινικέ έρευνες. Μετά αναφερθήκατε στον ρόλο των ε, τραπεζών είτε μιλάμε για εμπόριο ναρκωτικών είτε για έρευνες ε, της φορολογικής διοίκησης ε, οπότε βεβαίως δεν θα μπορούσα να σχολιάσω συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά στη χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα δεν έχω δει πρόβλημα για τη φορολογική διοίκηση να κάνει ελέγχους σε τράπεζες. Κάνουν ελέγχους, εξακολουθούν να κάνουν τους ελέγχους. Αλλά, ξέρετε, με την εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης ε, της οδηγίας ε, ε, για την αποταμίευση και την ανάγκη να αναφέρονται και τα κέρδη των επενδυτών και τα λοιπά, δημιουργούμε τις συνθήκες ε, ώστε οι τράπεζες ε, να ε, γίνουν πολύ πιο διάφανες και όπως σας είπα το τραπεζικό απόρριτο σύμφωνα με την ομοθεσία μας έχει τελειώσει. Δεν μπορεί καμία χώρα να αρνηθεί να ανταλλάξει πληροφορίες. Ε, επικαλούμε το τραπεζικό απόρριτο. Βεβαίως, ο συναδελφός μου, ο Μισελ Μπαρνιέ, κάνει πάρα πολλά στον τομέα των αλλαγών, στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η διαφάνεια είναι ένα στοιχείο αυτών των αλλαγών. Και γενικότερα βεβαίως της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και προς εκεί πάει το μέλλον. Οπότε νομίζω Πώς να κάλυψα. και ένα συγκεκριμένο ερώτημα που αφορούσε την Ιταλία. Πρέπει να σας πω ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν ερεύνησαν τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση και κατέληξαν ότι δεν υπήρξε παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Βασιζόμαστε βέβαια στην ανάλυση των υπηρεσιών μας γιατί οι επιπτώσεις μιας πιθανής παραβίασης θα κατέληγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε πολύ καλό παρελθόν όσες φορές προσφύγαμε εκεί, τις περισσότερες φορές κερδίσαμε τις υποθέσεις. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε. Απαντήσατε σε όλες μας τις ερωτήσεις ε, με ιδιαίτερη ακρίβεια και χαράξατε και μία φιλόδοξη πορεία. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας ε, ξαναδούμε ως ε, ομιλητή εδώ πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα σας καλώ όλους να φύγετε από την αίθουσα, εκτός ε, από τους συντονιστές, όσους θα συμμετέχουν στην εδρίαση των συντονιστών, η οποία θα γίνει και κλεισμένα των θυρών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Thank you